Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Καθίστε παρακαλώ. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε σήμερα τη δεύτερη μέρα αυτή των εργασιών μας. Το θέμα μας σήμερα, το πρώτο μας θέμα, είναι η πυρηνική ασφάλεια, διάσκεψη κορυφής δηλαδή για την πυρηνική ασφάλεια. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον ε, ειδικό σύμβουλο, τον κύριο σύμβουλο και ειδικό απεσταλμένο τη σήμερα εκπροσώπου, τον πρέσβη Γιάτσεκ Μπίλιτσα. Έχει ήδη συμμετάσχει σε διάφορες ε, συναντήσεις μας κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής εδώ στην Υποπιτροπή Σέντερ. Τον καλωσορίζω λοιπόν εδώ και χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλή μέρα αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, προκειμένου να σας ενημερώσω για την τέταρτη διάσκεψη πυρηνικής ασφάλειας που έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον 31 Μαρτίου με 1η Απριλίου του 2016. Όλη αυτή η διαδικασία της διάσκεψης αυτής κορυφής ξεκινάει από μια ομιλία του Πρόεδρου Ομπάμα στην Πράγα τον Απρίλιο του 2009 σχετικά με τα πυρηνικά ζητήματα και εκεί μίλησε για το όραμά του προκειμένου να έχουμε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα. Όμως χρόνος στην Πράγα ανακοίνωσε και μια νέα διεθνή προσπάθεια και παραθέτω προκειμένου να προστατευτούν όλα τα πυρηνικά υλικά, τα ευάλωτα πυρηνικά υλικά που βρίσκονται στον κόσμο μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο κύριος στόχος δηλαδή της πρωτοβουλίας αυτής είναι να μην μπορούν οι τρομοκράτες να έχουν πρόσβαση σε πυρηνικό υλικό. Συνεχίζεται η προσπάθεια αυτή ακόμα και τώρα. Προηγούμενες αντίστοιχες διασκέψεις είχαν γίνει στην Ουάσιγκτον το 2010, στη Σεούλ το 2012 και στην Χάγη το 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, ένας από τους τέσσερις διεθνείς οργανισμούς που προσεκλήθη στην ε, διάσκεψη αυτή κορυφής για την ασφάλεια από τα πυρηνικά του 2016 μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, τον Πανκιμούν, την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, τον Γενικό Διευθυντή Αμάνο και την Ιντερπολ που εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Στόκ. Ο πρόεδρο Τάσκ ήταν επικεφαλή τη Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είπατο εκπρόσωπο Μποκερίνη ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπησε έτσι τον πρόεδρο Γιούγκερ. Πάνω από 50 χώρες από ολόκληρο τον κόσμο και 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν προσκεκληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μεταξύ άλλων 35 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων που συζήτησαν για τους κινδύνους που απορρέουν από τα πυρηνικά αλλά και για άλλες μορφές τρομοκρατίας και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Το πρόγραμμα της μερούς αυτής της διάσκεψης αποτελεί το από ένα δείπνο στο Λευκό Οίκο, από την Ολομέλεια προκειμένου να συζητηθούν οι εθνικές δράσεις, ένα γεύμα εργασίας όσον αφορά τις διεθνείς και θεσμικές δράσεις για να ενισχυθεί η πυρηνική ασφάλεια και υπήρχε και συζήτηση πολιτικής πάνω σε ένα υποθετικό σενάριο τρομοκρατικής δράσης. Εκ παραλλήλου υπήρξαν, υπήρξε και μια διάσκεψη άλλη για τα πυρηνικά και μια άλλη πυρογνωμόνων όπου συμμετείχαν think tanks, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και κοινωνία των πολιτών. Όλες οι τάσεις συζητήθηκαν κατά το δίμερο αυτό συζητήσεων. Ο πρόεδρος Ομπάμα άκουσε πολλά θετικά μετά από την πρωτοβουλία αυτή του 2009 σε σχέση με απειλές από πυρηνική τρομοκρατία, τρομοκρατία κορπισμού, ραδιενέργειας και αυτό τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι διάφορες χώρες ετοίμασαν εκθέσεις πρόοδου για τα επιτεύγματά τους όσον αφορά την ασφάλεια από τα πυρηνικά και πώς ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί εμπλουτισμένο ουράνιο σε μη στρατιωτικούς σκοπούς και πώς θα ενισχυθεί η προστασία πυρηνικών υποδομών και υλικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δικιά της την πλευρά υπέβαλε μία έκθεση, ήταν το έγγραφο SWD 2016 198 98 που είναι έγγραφο εργασίας του προσωπικού και Έχω στη διάθεσή σας και κάποια αντίγραφα, αν θέλετε, και από το Joint Research Center, το κοινό ερευνητικό, την ερευνητική υπηρεσία. Είναι εδώ εκπρόσωποι που μπορούν να σας εξηγήσουν περισσότερα. Όταν άρχισε να ισχύει η σύμβαση για την φυσική προστασία από ε, πυρηνικό υλικό και υποδομές, αυτό ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα. Η αρχική σύμβαση είχε να κάνει μόνο με πυρηνικό υλικό το οποίο διακινείται διεθνώς. Όμως τώρα με τροπολογία καλύπτεται όλο το πυρηνικό υλικό, ακόμα και όταν αυτό διακινείται εσωτερικά, όταν πρόκειται για μη στρατιωτικού σκοπού και για αποθήκευσή του, όπως επίσης πρόκειται και για τις πυρηνικέ ε, υποδομές. Και είμαστε περήφανοι που όλε οι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Euratom έχουν κυρώσει την τροπολογία αυτή. Επίση, σύμφωνα με την πολιτική μα για την πρόθεση των διεθνών συμβάσεων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχει αναλάβει διπλωματική δράση προκειμένου να αρχίσει να ισχύει η συμφωνία αυτή. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει τα μάλα στο CPPNM και τι τροπολογίε του, προκειμένου να αρχίσει η τροπολογία αυτή να ισχύει από την 8η Μαου του 2016. Κατά τις συζητήσεις που έγιναν στη διάσκεψη, η τρομοκρατική απειλή κρίθηκε ότι αυξάνει, μετά μάλιστα από τις πρόσφατες επιθέσεις στο Βέλιο, την Τουρκία, το Πακιστάν και αλλού. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά μέσα, οι τεχνολογίες επικοινωνίες και ιδιαίτερα τα drones. Βάσει όλων αυτών λοιπόν συμφωνήσαμε ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των χωρών. Όσον αφορά τώρα τη διάδοση των πυρηνικών. Υπήρξαν επικρίσεις ε, στην ε, Βόρεια Κορέα εξαιτία τη προκλητική τη συμπεριφορά και απέναντι στη Ρωσία επίση που βασίζεται όλο και περισσότερο στα πυρηνικά όπλα και τον εξυγχρονισμό τους αποσύρθηκε από την ε, διάσκεψη η Ρωσία το 2014 σημειωτέων. Αναγνωρίστηκε επίσης η σημασία που έχει η συμφωνία με το Ιράν, JCPOA. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ρόλο κλειδί στη συμφωνία αυτή. Θέματα ασφάλειας από τα πυρηνικά ε, συζητήθηκαν επίσης γενικότερα για τους πυρηνικούς σταθμούς, για τους κινδύνους να υπάρξουν ε, ατυχήματα από τα οποία κινδυνεύουν γείτονες χώρες και για το θέμα της διαφάνειας. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πυρηνικός αφοπλισμός αναφέρθηκε επίσης από πολλούς ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των στόχων που έθεσε στην Πράγα ο πρόεδρος Ομπάμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν της διάσκεψης αυτής κορυφής του 2016 συμπεριλαμβάνει την δήλωση της διάσκεψης και πέντε προγράμματα δράσεις σε σχέση με το έργο των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, της Ιντερπολ, της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του, της πυρηνικής τρομοκρατίας και της ε, συνολικής εταιρικής σχέσης. Όλα αυτά υπάρχουν στο site www.nss2016.org. Ρόλο κλειδί παίζει η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας η οποία θα είναι υπεύθυνη να προχωρήσει το έργο της διάσκεψης αυτής στο μέλλον και να συμπεριλάβει και μια διεθνή διάσκεψη για την πυρηνική ασφάλεια που θα οργανώσει η διεθνής αυτή η υπηρεσία ατομικής ενέργειας στη Βιέννη 5 με 9 Δεκεμβρίου του 2016. Πολλές χώρες και οι αμφιτρίωνες Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην διάσκεψη αυτή σε υπουργικό επίπεδο. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν και πρόταση για μια τυπή ομάδα επαφής που θα συναντιέται στην Βιέννη μια φορά το χρόνο στο περιθώριο κατά πάσα πιθανότητα της διεθνούς αυτής διάσκεψης της CIA. Η άτυπη αυτή ομάδα θα είναι ανοιχτή σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Επιπλέον, η διάσκεψη έδωσε την ευκαιρία σε να λάβουν χώρα και άλλες ε, συναντήσεις και διμερείς διπλωματικές επαφές με τον πρόεδρο Τάσκα και την ε, κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ πολύ και με στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε ειδικοί απεσταλμένοι, κύριε Πρέσβη, ε, τα μέλη μας θα θέλανε να κάνουν κάποιες ερωτήσεις, να υποβάλουν κάποιες σκέψεις τους σε σχέση με τα όσα είπε ο πρέσβης κύριος Μπιλίτσα. Να ξεκινήσω εγώ με τις δικές μου ερωτήσεις. Πρώτον, είστε σίγουρος ότι ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή το 2009 και όχι το 2010. Εγώ αν θυμάμαι καλά Πράγα είχε λάβει χώρα ταυτόχρονα με την υπογραφή της START 2. Νομίζω ήταν Απρίλιο 2010. Το θυμάμαι για άλλους λόγους. Τι θυμάμαι αυτή τη συνάντηση της ε, Πράγας. Ε, δεύτερον, η αποχώρηση της ε, Ρωσίας από την πυρηνική πρωτοβουλία του 2014 ε, πράγματι ε, έλαβε χώρα και ακολουθήθηκε από άλλες αποφάσεις της Ρωσίας για την διεύρυνση και επέκταση των στρατηγικών της ε, ικανοτήτων, δυνατοτήτων. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό η, το φόρουμ της Βιέννης, το άτυπο φόρουμ της Βιέννης ε, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδεχόμενη πλατφόρμα για να επιστρέψει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ή υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Και πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ε, ασφάλεια των παλαιότερων πυρηνικών σταθμών. Ε, τι αποφάσεις έχουν λάβει διάφορες χώρες σε σχέση με αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Και σε ό,τι αφορά και την, το ενεργειακό μείγμα τους βέβαια. γιατί αυτό προφανώς ε, επηρεάζει την ε, δυνατότητα ε, μη κρατικών παραγόντων να φέρουν σε πέρα σε πυρηνικές επιθέσεις στο μέλλον. Άλλες ερωτήσεις. Okay, so, so please answer this. And... Oh, uh, sorry. Uh, pan poseł Mm, więc jeśli można, to mm, chciałem podziękować. Są zawsze ciekawe, ale... Ευχαριστώ για την, για την παρουσίασή σας. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Ε, η θέση της Ρωσίας και το ρωσικό ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η Ρωσία προφανώς δεν ήταν παρούσα σε αυτή τη συνάντηση, εντάξει. Αλλά να ρωτήσουμε για τον εαυτό μας, να ρωτηθούμε δηλαδή γιατί δεν ήταν παρούσα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Ρωσία επέλεξε πως δεν θα εφαρμόσει, δεν θα τηρήσει τους κανόνες που υπογράφηκαν στο παρελθόν ή αυτή τη στιγμή αναπτύσσει καινούριου τύπους πυρηνικού εξοπλισμού. Καινούριε πυρηνικές κεφαλές, για παράδειγμα ε, Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ανεξάρτητα το τι υπέγραψε τα προηγούμενα χρόνια η Ρωσία δοκιμάζει καινούρια όπλα. οι επωνομαζόμενες βρώμικες βόμβες, τα βρώμικα όπλα διασκορπισμού, ραδιενέργειας. Ε, φαντάζομαι ε, δεν ε, είναι εύκολο να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές. Αλλά σκάσιμο υλικό έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι τόσο δύσκολο κάποιος να αποκτήσει Τρίτον, η ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πριν από μερικές μέρες, οι Γερμανοί ζήτησαν από το Βέλγιο να κλείσει, να απενεργοποιήσει δύο αντιδραστήρες, διότι οι ειδικοί στη Γερμανία ισχυρίζονται ότι δεν είναι ασφαλής. πόσοι μη ασφαλείς πυρηνικοί αντιδραστές υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχετε στοιχεία, νούμερα. Πρόεδρος, ο κ. Κούζο Περμόη. Okay. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν ε, τον κύριο Μπιλίτσα για αυτές τις πληροφορίες. Να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες ε, ε, μη διάδοση η ε, και λοιπά. Όλες αυτέ οι βασικέ συμφωνίες κινδυνεύουν. Ε, εγώ ανησυχώ για την μεταφορά πυρηνικών όπλων, όπως για παράδειγμα από τι Ηνωμένε Πολιτείε στην Τουρκία. Ή όταν η Ρωσία μετακινεί τα σκάνερα στο στο Καλίνιγκραντ. Επίσης, ε, η απουσία του πυρηνικού προστασίου του Ισραήλ έλειπε, έλειψε από την ημερήσια διάταξη ε, της ε, Συνόδου Κορυφής, δεδομένης και της ομαλοποίησης κατάστασης με το Ιράν θα έπρεπε. Panie ambasadorze, może bardzo proszę o odpowiedź na e, ε, θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις κύριε Μπλίτσα. Ευχαριστώ πολύ για αυτές ε, τις ε, εχμηρές θα έλεγα ερωτήσεις. καταρχήν για τις ημερομηνίε. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε σε μια ομιλία του Πρόεδρου Ομπάμα στην Πράγα τον Απρίλιο του 2009. η, ομιλία και η ανακοίνωση έγινε τον Απρίλιο 2009. Εκεί είπε ότι η καινούρια πρωτοβουλία θα ξεκινήσει σε ένα χρόνο. Και πράγματι ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2010, έλαβε χώρα η πρώτη σύνοδος κορυφής στην Ουάσιγκτον. Έχω μπροστά μου την εικόνα του Ρόμπερτ Κουμπιέσκι του πρέσβη που αντικατέστησε την, τον πρόεδρο της Πολωνίας σε, ε, σε εκείνη τη συνοκορυφή, το θυμάμαι πολύ καλά. Αυτά σε ό,τι αφορά το χρόνο διάγραμμα της ημερομηνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία. Ας κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε τρία πράγματα. Πυρηνική ασφάλεια, η φυσική ασφάλεια ασφάλεια λειτουργίας, δύο πράγματα δηλαδή, και την μη διάδοση. Ε, το, ε, η φυσική ασφάλεια αφορά την ε, αποφυγή ατυχημάτων, όπως το Three Mile Island, το Chernobyl κλπ. Η ασφάλεια λειτουργίας αφορά την πρόληψη κακής χρήσης από τρομοκρατία κλπ. Και η μη διάδοση είναι η αποφυγή ε, απόκτησης ε, τέτοιων υλικών ή όπλων από χώρες ε, οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν ή απόκτηση περισσότερων όπλων από χώρες που ήδη έχουν. Τώρα, η Σύνοδος Κορυφής αφορά μόνο το δεύτερο από αυτά τα τρία πράγματα, την ασφάλεια λειτουργίας και την αποφυγή ε, τρομοκράτες να αποκτήσουν ε, τέτοιου είδους υλικά. Τώρα, στις συζητήσεις Βέβαια, ενεπλάξαν και άλλα ζητήματα, εθίγησαν και άλλα ζητήματα, όπως η παραβίαση του memorandum της Βουδαπέσης από τη Ρωσία κλπ. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει ότι αποκτά καινούριους ο, ο, καινούς τύπους όπλων. Τώρα, αν αυτό παραβαίνει τις συμφωνίες ή όχι, οι Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι παραβαίνει η Ρωσία τη συμφωνία και ιδιαίτερα τη συμφωνία, πολύ σημαντική συμφωνία για την Ευρώπη. Και αυτό παντά εν μέρει και στην ερώτηση του κ. Ζέμκα, την INF για τις ε, πυρηνικές ε, ε, δυνάμεις μέσου βεληνικού στην Ευρώπη που ε, αφορά ε, βελνικές από 500 έως 5.500 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ σημαντική για την ασφάλεια της Ευρώπης γιατί έχουμε μια ολόκληρη κατηγορία πυρηνικών όπλων τα οποία έχουν πλέον αποσυρθεί από την Ευρώπη και έχουν καταστραφεί με επαλήθευση περίπου 3.000 τέτοιου είδους ε, κεφαλές. Οπότε οι ισχυρισμοί περί παραβίασης της συνθήκης INF είναι πολύ σημαντικοί και βαρύνουν. Ελπίζουμε ότι η συνθήκη θα συνεχίσει να λειτουργεί με επαληθεύσεις και δεν θα καταρρέψει όπως άλλες συνθήκες στο παρελθόν. Και εδώ απαντώ την ερώτηση του, της Προέδρου πού μπορούν να συζητηθούν αυτά με τη Ρωσία. Η Βιέννη, ε, στη Βιέννη συζητούνται θέματα ελέγχου συμβατικών όπλων και εκεί η Ρωσία ανέστηλε τη συνθήκη, τη CFE, περί ε, ε, συμβατικών όπλων στην Ευρώπη, ε, αλλά εκεί στη Βιέννη συζητούνται θέματα συμβατικών ε, όπλων. Και βέβαια και μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης, όπως για παράδειγμα αμοιβαία ανακοίνωση ε, ε, ασκήσεων κλπ. Ε, καθώς επίσης και η συνθήκη περιπερτήσεων. Ε, είναι πιο συμβατικά θέματα λοιπόν αυτά που συζητούνται στην Βιέννη. Οι στρατηγικές συζητήσεις ε, γίνονται κυρίως διμερώς μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Παρόλο ότι επισήμως τυπικά σύμφωνα με τη συνθήκη INF, άλλες χώρες όπως η Ουκρανία και η Λευκορωσία, που είναι διάδοχες χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, επίσης εμπλέκονται. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας και της ασφάλειας ε, πυρηνικών σταθμών, ε, φυσική και λειτουργική ασφάλεια, ε, και εδώ έχουμε διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η, ασφάλεια σε ό,τι αφορά την πρόληψη ατυχημάτων ε, είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνονται stress test σε όλα τα ε, πυρηνικά εργοστάσια και πυρηνικού σταθμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Σε ό,τι διαφορά την ε, φυσική ασφάλεια, εξακολουθεί να είναι θέμα της αρμοδιότητας των κρατών μελών, το, το, το, το, safety δηλαδή. Τώρα, η ασφάλεια ραδιενεργών πηγών που πολύ συχνά ε, βρίσκονται πιο εκτεθειμένες όπως για παράδειγμα σε νοσοκομεία και δυστυχώς υπάρχουν ε, δεκάδες, ε, μα, χιλιάδες τέτοιου τύπου πηγές ραδιενέργειας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βρώμικες βόμβες. Οι δυνατότητες μιας τρομοκρατικής οργάνωσης να είναι αποκτήσει μια πυρηνική κεφαλή, λειτουργική πυρηνική κεφαλή, να την φτάσει, να τη φτιάξει από κλαπέν υλικό είναι πολύ χαμηλή. Έτσι, πολύ χαμηλή πιθανότητα. Όμως, μια βρώμικη βόμβα είναι τελείως διαφορετική, γιατί εκεί τα εκρηκτικά είναι συμβατικά. Ε, ο αριθμό των θυμάτων από μια τέτοια επίθεση θα είναι αρκετά περιορισμένο. Όμω, ο πανικό ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος θα είναι τρομακτικός. Δημοσιεύτηκε ένα άρθρο που έλεγε «Ας φανταστούμε τι θα γινόταν αν οι ε, ε εκρήξεις στο Ζάβεντεμ ήταν δρόμικες βόμβες ε, με ραδιενεργό υλικό και χρειαζόταν μετά να καθαρίσουμε το αεροδρόμιο». Ε, τόφορα η πρωτοβουλία NSS της ε, ε, Συνόδου για την πυρηνική ασφάλεια. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε την Ρωσία. Αντικειμενικά μιλώντας, ένας αριθμός, μεγάλος αριθμός από αυτές τις ενδεχόμενες πηγές ε, βρίσκεται στην επικράτηση της Ρωσίας και είναι κρίμα που η Ρωσία αποσύρθηκε το 2014 λέγοντας, ισχυριζόμενοι ε, επισήμως ότι ε, ε, οι, οι σύνοδοι αυτές ε, δεν συμπεριλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Τους πήρε τέσσερα χρόνια να το καταλάβουν αυτό. Ε, λέγανε ότι καλούνται 50 χώρες αντί για 200. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν πρόσχημα πλευράς της Ρωσίας. Όμως υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες όπου μπορεί και θα έπρεπε να συνεχιστεί η συνεργασία με τη Ρωσία. Ένα, μία από αυτές τις πλατφόρμες είναι GICNT που είναι ε, η παγκόσμια ε, πρωτοβουλία ε, όπου συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες. Ένα άλλο φόρουμ όπου μπορεί να λάβει χώρα συνεργασία για την ενίσχυση της ασφάλειας και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου είναι, και εδώ απαντώ στην ερώτηση του Ισπανού βουλευτή, ε, η Επιτροπή 1540 στη Νέα Υόρκη που εφαρμόζει το ψήφισμα του ΟΗΕ 1540. Ψήφισμα ε, επιτροπή η οποία αναδομείται φέτος με την, υπό την προεδρία του Ισπανού πρέσβη. Ε, πρόκειται για ένα ψήφισμα υποχρεωτικής εφαρμογής για όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ ε, και υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ποινικοποιήσουν ε, τις ε, δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών όπλων. Ε, θα πρέπει δηλαδή αυτό να αποτελεί αδίκημα και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ενημερώσουν για το πώς το έπρεξαν αυτό. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει και οικονομικά αλλά και με εμπειρογνώμονες για να ενισχυθούν οι, τα σύνορα στις γειτονικές μας χώρες έτσι ώστε ε, να εντοπίζονται στα σύνορα ε, πυρηνικές ουσίες, ραδιενεργές ουσίες. Ξέρετε, πολύ συχνά ε, ε, περνώντας τα σύνορα με ένα αυτοκίνητο ε, κανείς επιβραδύνει και περνάει από τους ε, φρουρούς, ε, αλλά στην πραγματικότητα δεν, δεν ελέγχεται καθόλου. Γίνεται μια μέτρηση ραδιενέργειας και εκεί φαίνεται και το ίδιο σημαίνει και στα φορτηγά. Είναι ένας έλεγχος ο οποίος γίνεται με τρόπο αόρατο, γιατί αόρατη είναι και η ραδιενέργεια, αλλά λαμβάνει χώρα και η Υπηρεσία Εξωτερικής αλλά και το Κοινό Κέντρο Ερευνών και η Euratom στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκονται πολύ ενεργά σε αυτό. Τέλος, το θέμα του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής. Οι συζητήσεις για την ε, ε, για την, να καταστεί το Ισραήλ ελεύθερο ε, ε, για τη ζώνη μάλλον που θα είναι ελεύθερη από όπλα μαζικής καταστροφής συζητήθηκε αλλά δεν υιοθετήθηκε ένα τελικό έγγραφο. Η ίδια η συμφωνία υπάρχει ισχύει και ελπίζουμε θα ενισχυθεί στον επόμενο κύκλο που θα ξεκινήσει του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Μετά από αυτά που είπατε, είχατε την απάντησή σας ή θέλετε να σχολιάσετε παρετέρω. οι δύο ομιλητές που υπέβαλαν ερωτήσεις. Όχι, εντάξει. Καλώς τότε. Έτσι ολοκληρώνεται αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Εντάξει, το ενδιαφέρον είναι αυτό που είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πρέσβη, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Εδώ κλείνει το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη, αλλά μπορείτε να παραμείνετε μαζί μας, γιατί θα περάσουμε ευθύ αμέσω στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αντιπροσωπείας μας που πήγε στο Νόρτβέικ και περάσαμε εκεί μια ολόκληρη μέρα. Σας ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, Κυρίες και κύριοι, πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Δεν είναι βέβαια ουσίας. Συμμετείχαν διάφοροι ευρωβουλευτές στην επίσκεψη αυτή. Δεν είναι όλοι εδώ παρόντες. Οπότε νομίζω ότι εγώ θα πρέπει να σας ενημερώσω για την επίσκεψή μας αυτή στο Νόρτβέικ. Ως ε, ήθιστε, η ΣΕΝΤΕ, η Επιτροπή μας δηλαδή, πήγε ε, στο, στην έδρα, στο στρατηγείο της ε, υπηρεσίας αυτής. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψή μας, πρέπει να σας πω. Περάσαμε μια ολόκληρη μέρα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και στην επίσκεψη αυτή μα συνόδευσε προσωπικό ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και επαγγελματικών προσόντων. Μπορέσαμε έτσι να παρακολουθήσουμε την αξιολόγηση των ικανοτήτων του κέντρου αυτού, την αριστεία του. Και αυτά ξέροντας ότι με την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Διαστήματος ε, γίνονται διαγωνισμοί, δημιουργούνται κονσόρσια, προκειμένου η υπηρεσία αυτή να πετύχει τους ε, στόχους της, χρησιμοποιώντας τις σωστές διαδικασίες ανταγωνισμού όσον αφορά το διάστημα. Μπορέσαμε επίσης να επισκεφθούμε διάφορα εργαστήρια εκεί. Είδαμε επίσης να γίνονται δοκιμές με δορυφόρους για την ακρίβειά τους. Είδαμε τεχνολογικά δηλαδή πόσο ακριβείς μπορούν να είναι οι δορυφόροι. Κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Είδαμε λοιπόν στα εργαστήρια πώς εργάζονται και τι είναι διαθέσιμο. Όλα αυτά χάρη στην ευγενή καλοσύνη του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε και την λειτουργική δυνατότητα ε, του κέντρου εκεί. Μέτρα ασφάλειας, πώς λειτουργεί δηλαδή αυτό το κέντρο. Και η επίσκεψη αυτή ήταν μία από τις πιο σημαντικές. Βέβαια έλαβε χώρο λίγο πριν, έλαβε χώρο λίγο πριν εγκρίνει η ΑΦΕΤ την έκθεση για τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής όσον αφορά το διάστημα. Ο εισηγητής εδώ στη ΣΕΝΤΕ δύο φορές ήρθε να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. παρουσιάσαμε και εμείς τις δικές μας ιδέες, υπήρξαν πολλές τροπολογίες και τελικά εγκρίθηκε η έκθεση αυτή. Οι ευρωπαϊκές χώρες μέλη και το προσωπικά της ESA θεωρούν ότι πρόκειται για ακρογωνίο λίθο που καλύπτει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαστήματος. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλο τη γραμματεία, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος που οργάνωσε μαζί μας την ε, επίσκεψη αυτή. Τώρα, αν οι ευρωβουλευτές θέλουν να σχολιάσουν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yeah, okay. So we are satisfied. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στο ταξίδι μας αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς που βάλατε το θέμα αυτό στην μερική διάταξη της Υποπιτροπής μας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να συζητάμε για τέτοιου είδους τεχνολογία εδώ, είναι πιο εύκολο, πιο απτό όταν κανείς πηγαίνει επί τόπου. Τα τεχνολογικά αυτά κέντρα, σαν και αυτό που επισκεφθήκαμε, υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Αλλά αυτό ήταν ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος. Και ισχύει και για άλλες επιτροπές, οπότε σε κάποια άλλη ευκαιρία να το συζητήσουμε εδώ στην υποπιτροπή μας. Πρόεδρος, ναι. Νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σας, κύριε Στρογεύσκη για τα αποτελέσματα της επίσκεψης αυτής και ευχαριστώ και εγώ για τα σχόλια. Ίσως το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς να επανέλθουμε εδώ. Γιατί το διαστημικό πρόγραμμα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βέβαια και αυτό από πολλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Με την ΑΦΕΤ ε, υπάρχει κοινή ακρόαση που θα οργανώσουμε. Θα συζητήσουμε την προστασία του κυβερνοχώρου σε λίγο και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις απειλές. Στις 10.30 θα αρχίσουμε και πάλι, ακριβώς.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 No, Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 parler à... Donc 1, 2, 3, 4, ok, et, et, et,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 boy comment Υπότιτλοι AUTHORWAVE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

Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της κυρίας Φωτίγα και μου του ιδίου κήρυσω την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η οποία μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Και από τα γραφεία μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι συνάδελφοι και εκτός. Έχουμε λοιπόν σήμερα την ακρόαση αυτή για τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την προστασία της Ευρώπης και των πολιτών της. Δεν υπάρχει μόνο το στρατιωτικό σκέλος, είναι ένα γενικότερο θέμα που αφορά την κοινή μας πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος μπορεί να διακόψει την οικονομική ανάπτυξη, για παράδειγμα. Υπάρχουν ένα σωρό κίνδυνοι που απορρέουν από τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Κινδυνεύουν οι πυρηνικοί σταθμοί, για παράδειγμα. Οι απειλές οι ηλεκτρονικές είναι πάρα πολλές και αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Είναι και πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εκπονήσουμε τις κατάλληλες πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την απειλή αυτή του ηλεκτρονικού πολέμου. Πολλές χώρες ετοιμάζονται για συγκρούσεις στον κυβερνοχώρο και οι ικανότητές μας πρέπει να αναπτυχθούν παρετέρω για να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Η αντοχή μας πρέπει να ενισχυθεί επίσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε ακόμα περισσότερο ώστε να αναπτύξουμε τα κατάλληλα δίκτυα ηλεκτρονικής ασφάλειας. Πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπαθειές μας. Σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Ε, δυστυχώς πολλές φορές δεν υπάρχει συνοχή στην προσέγγισή μας και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με ανησυχεί. Έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά πάντως στο τομέα της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ήδη από το 2014. Ξακολουθεί όμως να υπάρχει κάποια αντίσταση από ορισμένε χώρες μέλη για να συνεργαστούν αμοιβαία υπέρ της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τι λοιπόν μπορεί να γίνει για να ενισχύσουμε την δυνατότητα αντίστασής μας Πολλά μπορούν να γίνουν σε διπλωματικό επίπεδο πρώτα απ' όλα. Έπειτα να υπάρχουν κανόνες, κανόνες συγκρίσιμοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς για να υπάρξει μια αμοιβαία κατανόηση των κανόνων και της συμπεριφορά στον κυβερνοχώρο. Οι ειδικοί λοιπόν μπορούν να μας πούν τι προτείνουν να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να συνεργαστεί στενότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ προκειμένου να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας παραπάνω. Υπάρχουν πολλά μέσα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλον και πολλά έχουμε να μάθουμε από το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ κάνει πολλή δουλειά όσον αφορά την προστασία του κυβερνοχώρου. Τέλος, Θέλω να υπογραμμίσω ότι πρέπει να αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής η προστασία του κυβερνοχώρου. Οι εξελέξεις προχωράνε γρήγορα στο εξωτερικό. Επιπλέον, πρέπει να μάθουμε και περισσότερα για τους υβριδικούς πολέμους. Είναι πεποίθησή μου ότι πρέπει να ξαναδεί την πολιτική της ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει μια πιο πλήρη αντίληψη για την έννοια της ε, ηλεκτρονικής ασφάλειας, να λάβει υπόψη όλες τις ε, διαστάσεις, την τρομοκρατία για παράδειγμα και όχι μόνο τις συμβατικές απειλές. Το νέο πεδίο στον κυβερνοχώρο απαιτεί περισσότερη συνεργασία. μεταξύ διαφορετικών παραγόντων και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο χωρών μελών. Οι απειλές ηλεκτρονικές δεν σταματούν στα σύνορά μας. Γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών και παρετέρω ανάπτυξη της ικανότητάς μας και συνεργασία. Ελπίζω όλοι να το ανταλαμβάνονται έχουμε νομίζω αρκετές εμπειρίες για να ξέρουμε ότι υπάρχει ανησυχία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φωτίγκα που είναι πρόεδρος της ε, ΣΕΝΤΕ και μετά θα ακούσουμε τους ειδικού μας. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ναι, πράγματι, όπως ε, τα είπατε, θα έλεγα ότι το καμπανάκι του συναγερμού έχει χτυπήσει. Τώρα έχουμε περισσότερη εμπειρία. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος είναι κάτι που απειλεί την ηλεκτρονική μας ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά θα σας παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε την κυρία Χέλη Τίρμα Κλάρ από την EAS, η οποία θα μας παρουσιάσει το τι γίνεται όσον αφορά το συντονισμό για την ηλεκτρονική ασφάλεια. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι θεσμικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η EAS είναι και το αρμόδιο όργανο. Έχουμε μετά τον κύριο Steve Purser, ο οποίος θα μας ε, μιλήσει πιο πολύ για τις ειδικέ και τις βιομηχανικές πτυχές του ζητήματος. Εκπροσωπεί την ΕΝΙΣΑ. Είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και εφόσον δεν πρόκειται μόνο για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, θα μας μιλήσει και για την διάσταση του ΝΑΤΟ. Εξού και έχουμε και τον κύριο Κρίστιαν Μάρκ Λίφλεντερ, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΝΑΤΟ αυτός. Μετά λοιπόν από αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις που θα ακούσουμε, θα ακολουθήσει η συζήτηση. Λοιπόν, πρώτα η κυρία Τύρμα Κλάρ, μετά ο κύριος Πέρσερ και στη συνέχεια ο κύριος Λίφλεντερ. Μετά θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις και ενδεχομένω και δεύτερο γύρο. Λοιπόν, έχετε το λόγο κυρία Τίρμα Κλάρ. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι το ζήτημα αυτό αποκτά όλο και μεγαλύτερη πολιτική σπουδαιότητα. Αποτελεί ζήτημα που θα μας απασχολεί στο μέλλον. Εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και είμαι τμήματάρχης ενός μικρού τμήματος που ασχολείται με την διπλωματία, τις ξένες σχέσεις στον κυβερνοχώρο και την πολιτική άμυνας. Να ξεκινήσουμε τα ζητήματα κυβερνοδιπλωματίας. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Μπρόκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ρόλο παγκοσμίω όσον αφορά τη συζήτηση περί προτύπων στον κυβερνοχώρο και πώς μπορούμε να αποφύγουμε έναν μεγάλο κυβερνοπόλεμο στο μέλλον. Θα ήθελα να σας πω ότι οι προσπάθειες αποφυγής ε, μεγάλης διαμάχης στον κυβερνοχώρο έχει ξεκινήσει ήδη μετά από τις επιθέσεις του 2007 στην Εσθονία, η οποία έθεσε το θέμα στον ΟΣΑ, στα Ηνωμένα Έθνη, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πίεσε τους μεγάλους ε, οργανισμούς να ασχοληθούν με, την, ε, με μέτρα αποφυγής κλιμάξης ε, διαμαχών στον κυβερνό χώρο. Όπως τα λέμε στη διπλωματία, είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πολιτικής εμπιστοσύνης, τα οποία πραγματοποιούνται δυνάμεις συμφωνιών μεταξύ των μεγάλων κυβερνήσεων, ώστε να αποφύγουμε ορισμένες διαμάχες ορισμένους τομείς. Οι εργασίε αυτέ έχουν προωθηθεί στον ΟΣΑ με την υποστήριξη των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του προσωπικού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκολύνοντας εκεί το συντονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση Και ήδη από το 2013 είχαμε τα πρώτα μέτρα τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ 24 ε, χωρών του ΟΣΑ. Το 2016, το Φεβρουάριο, είχαμε το δεύτερο σύνολο μέτρων ε, οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμφωνήθηκαν για την ασφαλή στον χώρο. Τα πρώτα μέτρα ονομαστικά μέτρα διαφάνειας περιλαμβάναν σε σημεία επαφής, τις κοινέ εκδηλώσεις, την κοινή χρήση πληροφοριών για τις διαφορές πολιτικές και το δεύτερο σύνολο μέτρων ονομάζεται μέτρα διαφάνειας. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία δηλαδή μεταξύ των χωρών και πιο καλή κατανόηση των ε, εκατέρωθων προθέσεων. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη ε, είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή αποφυγή ε, ε, διενέξεων στον τομέα αυτών. Έχει πιέσει το ζήτημα να προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός της ευρωατλαντικής περιοχής. Το Μάρτιο διοργανώσαμε ένα σεμινάριο για τα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης στην περιοχή ΑΣΕΑΝ στο σχετικό φόρουμ. Ε, ε, το Περιφερειακό Φόρουμ του ΑΣΕΑΝ ε, έχει μέλη τις μεγάλες χώρες της Ασίας, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται και οι περισσότερες ασιατικές χώρες. Προσπαθούμε λοιπόν να καλύψουμε τον τομέα της οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τρόπο τέτοιο ώστε να ενημερώνονται και οι υπόλοιπε χώρες εκτός της Ευρωατλαντικής περιοχής. Όσον αφορά τα πρότυπα, Αυτά διαφέρουν από τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, τα οποία είναι περισσότερο πολιτικέ συμφωνίε μεταξύ κυβερνήσεων. Και αυτή τη λίστα μέτρων πρέπει να προσυπογράψουν ε, όλε οι χώρε και διάφοροι οργανισμοί όπω ε, ο ΣΑ τα πρότυπα όμως ε, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι μια ευρύτερη διαδικασία και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία στον ΟΗΟ ε, με διαφορούς κυβερνητού ε, εκπροσώπους οι οποίοι συνέρχονται σε μια ομάδα η οποία έχει εκπονήσει πολλές εκθέσεις περί συμφωνιών μεταξύ των διαφορών κυβερνήσεων για το πώ αυτέ οι κυβερνήσει θα συμπεριφερθούν ώστε να αποφύγουν μέγιστέ διενέξει και πώ θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στο τι ε, είναι πιο πιθανό να δεχθεί επίθεση και τι όχι σε περίπτωση διένεξη στον κυβερνοχώρο. Οι ομάδες ε, απόκρισης ε, σε περίπτωση επιγόντων περιστατικών στους υπολογιστές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί και είναι μια καλή αφετηρία δήλωση των ουδέτερων ζωνών στον κυβερνοχώρο. Ε, όπως έχουμε τις ουδέτερες ζώνες, τις, ε, κλασικές ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν επιτιθέμεθα σε νοσοκομεία ή σε ουδέτερες περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετέχει σε αυτή την ομάδα, η οποία είναι άτυπη στον ΟΗΕ, αλλά κάποια κράτη-μέλη εκπροσωπούν τις γενικές απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Μέλη αυτής της ομάδας του ΟΗΕ έχουν έρθει στις Βρυξέλλες, στην ομάδα εργασίας ε, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο Συμβούλιο, ενημερώνοντας τα άλλα κράτη-μέλη. Και έτσι έχει γίνει και ιστορικά μια συζήτηση ε, στο Συμβούλιο με τα κράτη-μέλη για τη διαδικασία πρότυπων ε, στα, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο χώρο στα ΕΟΝΟΙΕ. Υπάρχει και άλλο ένα διπλωματικό στοιχείο πέραν των προτύπων που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και που προσθέτει αξία στη συνολική σταθερότητα στον χώρο παγκοσμίω. Είναι η αύξηση της γενικής ετοιμότητας των χωρών παγκοσμίω ώστε να αντιμετωπίζουν τις απειλές στον χώρο. όπου επενδύει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προγράμματα ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών, για να βοηθήσει τι αναδυόμενε χώρε και οικονομίε, για να δημιουργήσει τη βασική νομοθεσία και να λάβει τα βασικά τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να μπορεί να αποκριθεί, να αποκριθεί σε τέτοιες επιθέσεις διότι η πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική ε, σήμερα σε πολλές ε, αφρικανικές χώρες δεν υπάρχει καν άνθρωπος ε, ως επαφή με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει κανείς σε περίπτωση επίθεσης οπότε πρέπει να αναπτύξουμε το όλο δίκτυο επαφών και να αυξήσουμε τις δυνατότητες ε, που υπάρχουν ε, ε, το προσωπικό και τα μέσα. Κατά τις επιθέσεις στην Εσθονία, οι επιθέσεις αυτές ήταν της μορφής άρνησης εξυπηρέτησης. Μιλάμε για ψηφιακούς στρατιώτες που επιτέθηκαν σε τράπεζες και σε online υπηρεσίες της εσθονικής κυβέρνησης το 2007 κατά την πολιτική προεκλογική εκστρατεία τότε. Η εστονική κυβέρνηση κάλεσε όλες τις χώρες ε, και τις είπα να κλείσουν τα spotnet αυτά τα οποία προκάλεσαν τις απειλές, ε, προκάλεσαν τις επιθέσεις, αλλά σε ορισμένε περιπτώσει αυτό δεν ήταν δυνατόν και δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν τι επιθέσει. Και όπω μα έχουν πει, κάποιοι από αυτά τα σπότνετ του χτυπούν ακόμα και σήμερα, ε, δέκα χρόνια σχεδόν μετά από τι επιθέσει του 2007 διότι δεν ελέγχονται αυτές οι περιοχές. Κανείς δεν είναι υπεύθυνο ε, για τι υπηρεσίε στον κυβερνοχώρο εκεί. Οπότε προσπαθ... αυτή η ανάγκη ευαισθητοποίηση και εκτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό. Όχι μόνο για αυτού, αλλά και για εμά. γιατί όταν μα χτυπούν πρέπει και εμεί να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιον, να συνομιλήσουμε με κάποιον σε αυτές τι χώρες. Να σας μιλήσω τώρα για την άμυνα στον κυβερνοχώρο και για το τι κάνουμε εκεί. Έχουμε το πλαίσιο πολιτικής το οποίο συμφωνήθηκε και υιοθετήθηκε το 2014 με κάποιους στόχους. Όπως γνωρίζετε, ε, η CSDP ε, ε, είναι το πλαίσιο βάσει το οποίο ορίζονται όλα αυτά και οι αποστολές και οι επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφαλείας και πολιτικής άμυνας είναι το πλαίσιο αυτό Πέντε είναι οι στόχοι. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των ε, κρατών μελών στο πλαίσιο του CSDP. Δεύτερον, ενίσχυση των δικτύων προστασίας που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, προώθηση μη στρατιωτικής και στρατιωτικής συνεργασίας και εξέβρεση συνεργειών στο πλαίσιο των πολιτικών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κυβερνό χώρο, εκπαίδευση και κατάρτιση και ασκήσεις και τέλος ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ο συνάδελφος από το ΝΑΤΟ πιθανώς θα σας αναφέρει και αυτός ότι είχαμε μια μεγάλη επιτυχία τον Φεβρουάριο με την υπογραφή της Συμφωνίας Ανταλλαγής Πληροφοριών ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Είναι μια συμφωνία που ετοιμαζόταν για 13 χρόνια ε, υπογράφηκε λοιπόν για την ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών. Επίσης έχουν γίνει καλές προσπάθειες ε, για διαβουλεύσεις ε, μεταξύ προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την, ασφάλεια, την άμυνα στον κυβερνό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας έχουν αναθέσει τα κράτη-μέλη πρώτα απ' όλα να εστιαστούμε στην προστασία των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό αποτελεί τώρα προτεραιότητα. Επίσης κάνουμε πολλή δουλειά με τα κρατη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Άμυνας που έχει και την ομάδα έργου με τα κράτη-μέλη για τις ε, πιο μακροχρόνια οικοδόμηση ικανοτήτων για την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Επίσης ε, δραστηριοποιούμαστε στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις ασκήσεις Προσπαθούμε να απλουστεύσουμε όλα τα στοιχεία και να τα συμπεριλάβουμε και σε άλλες ασκήσεις που δεν ε, είχαν τέτοια διάσταση ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρωτήτερα. Και τώρα διαπραγματευόμαστε με την ΕΝΙΣΑ και με την ε, Cyber Europe ε, που είναι μια μη στρατιωτική άσκηση των κρατών μελών. Αλλά φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΗΣΑ θα είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει τι ακριβώς αρμοδιότητα έχει στον τομέα. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες. Το βασικό εμπόδιο όσον αφορά την άμυνα στον χώρο για εμάς είναι η έλλειψη πόρων. Οι πόροι μας είναι ανεπαρκείς, ε, τόσο ανθρώπινοι πόροι, τόσο όσο και ηλικοί και με το 5% περικοπές όλοι αυτοί είναι οι τομείς όπως ο κυβερνοχώρος έχουν υποστεί περισσότερες ε, ελλείψεις από ότι άλλες, ε, άλλοι τομείς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε βέβαια με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε. Επιτρέψτε μου να κλείσω με την δήλωση ότι δεν είμαστε μόνο εμείς ε, εδώ, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Μπροκ, είναι μια παγκόσμια, ε, ολιστική προσπάθεια αυτή στον κυβερνοχώρο και η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζεται στην ενίσχυση των ε, σχέσεών της στον κυβερνοχώρο με βασικούς εταίρους. Έχουμε ξεκινήσει διαλόγους για το θέμα αυτό με τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα. Πρόκειται για διαλόγους όπου συμμετέχει ο ΙΕΣ, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Έχουμε ορίσει την ατζέντα μαζί με τα κράτη-μέλη και μαζί με τους συναδέλφους μας από τα θεσμικά όργανα και αυτή η διαλογή μας βοήθησαν να θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε αυτές τις σχέσεις και τη συνεργασία στον τομέα του κυβερνοχώρου με άλλα μέρη του κόσμου. Ακόμη και με διαφορετικέ νοοτροπίε χώρε όπω η Κίνα έχουμε σημειώσει αρκετά καλή πρόοδο ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε για τη ε, δημιουργία των προτύπων και ούτω καθεξή. Επίση, πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε ότι οι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν και σε άλλε χώρε απαραίτητα. Οπότε αυτό είναι ο ρόλο μα και ευθύνη μα να αναφέρουμε την ε, εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για την ελευθερία του λόγου online. Έτσι με του διαλόγους αυτού για τον κυβερνοχώρο μπορούμε να επηρεάσουμε του εταίρου μα προ αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν και πολλέ μη στρατιωτικέ πτυχέ. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή μέσω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθηθεί από αυτέ. Και υπάρχουν και διάφορε εσωτερικές πτυχέ, που μερικέ φορέ είναι πιο σημαντικέ από τις εξωτερικές πολιτικές τη πολιτική ε, άμυνα, ώστε να αντισταθούμε σε έναν κυβερνοπόλεμο εντό τη Ευρωπαϊκής ε, όταν εξετάζει κανεί την ετοιμότητα των χωρών, παρατηρεί ότι υπάρχει, σχηματίζεται μια πυραμίδα. Θα πρέπει να υπάρχουν και μη στρατιωτικά στοιχεία, ε, μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων, μη στρατιωτική απόκριση ε, και κάποιες δομές μη στρατιωτικές για την αντίσταση σε τέτοιες επιθέσεις. Διότι όταν συμβαίνουν τέτοιες επιθέσεις πλήττουν κρίσιμες υποδομές, δίκτυα ενέργειας, ενδεχομένως δίκτυα ίδρυυσης, τράπεζες, και άλλες ε, εταιρείε που βασίζονται για τις εργασίες τους στον κυβερνό χώρο. Οπότε ακόμη και ο καλύτερος στρατός του κόσμου δεν θα μπορέσει να νικήσει ένα τέτοιο πόλεμο. Χρειάζεται λοιπόν μια προσπάθεια της συνολικής κυβέρνησης ε, που σημαίνει περίπου 85% μη στρατιωτικέ προσπάθειες και μετά μπορούν να παρέμβουν και οι στρατιωτικές δυνάμεις. Ε, κλείνω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τυρμακλάρ, ο κύριος Πέρσερ από την Ενίσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως θα μπορούσαμε να προβάλλουμε την παρουσίαση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. ε, ασύνηθες το κοινό για μας σήμερα, αλλά σίγουρα θα αλλάξει αυτό, ε, διότι το φαινόμενο της πολιτικοστατιωτικής συνεργασίας γίνεται όλο και πιο τακτικό και συχνό. Ας ξεκινήσω μιλώντας λίγο για την ΕΝΙΣΑ, πώς λειτουργούμε, ποιο είναι το λειτουργικό μας μοντέλο και μετά θα εστιάσω σε δύο βασικές ε, ε, πτυχές της συνεργασίας, CIIP και ανταλλαγή πληροφοριών το 90% περίπου των όσων κάνει η Ενίσα δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την παρουσίαση, οπότε αν θέλετε να έχετε πλήρη ενημέρωση, παρακαλώ ε, ελάτε σε επαφή μαζί μου. Ποια είναι η Ενίσα λοιπόν. Η Ενίσα δημιουργήθηκε, συστάθηκε το 2004 και η αρχική μας εντολή ανανεώθηκε το 2013. Είμαστε μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πυλώνα 1 δηλαδή για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς. Είμαστε κανονιστική υπηρεσία, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε την δυνατότητα να διαφωνούμε με, τους, ε, με τα θεσμικά όργανα, προσπαθούμε να μην το κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως ε, ε, ελέγχουμε την δράση των θεσμικών οργάνων, δίνουμε συμβουλές με ανεξάρτητο τρόπο σε ό,τι διαφορά τον ρόλο μας. Ε, το πιο ενδιαφέρον ίσως είναι ότι στην εντολή μας έχουμε την αποστολή ε, ε, να γεφυρώσουμε τον ιδιωτικό με το δημόσιο τομέα και το κάνουμε σε μεγάλο βαθμό. Ε, η ΕΝΙΣΑ ε, έχει 84 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων 55 είναι στη στο λειτουργικό κομμάτι, το, του οποίου ε, είμαι επικεφαλής. Έχουμε ένα προεπιλογισμό 10 εκατομμυρίων, ε, ελάχιστα σε σχέση με το μέγεθος του, προ, προβλήματος και ο προεπιλογισμός δεν έχει αυξηθεί και πολύ τα τελευταία χρόνια, ελάχιστα, ενώ το πρόβλημα και γενικότερα το ζήτημα έχει διαβρυνθεί, έχει ε, υποκτήσει εκρηκτικές ε, διαστάσεις. Έχουμε μια... Ο ειδικό μου προπολογισμό είναι 2 εκατομμύρια μόνο, για να το ξέρετε. Τώρα, πώς λειτουργούμε. Ε, κάνουμε ε, τα πάντα μέσω κοινοτήτων λειτουργίας. Ε, είναι όλο το προσωπικό μου, είναι εμπειρογνώμονες, είμαι περήφανη για αυτούς, αλλά ε, τη δική μας εμπειρογνωμοσύνη την συμπληρώνουμε με εμπειρογνωμοσύνη από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή συνδυάζουμε το δικό μας έργο μαζί με τους ανθρώπους που λειτουργούν στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε κοινότητες λοιπόν, μάλλον ε, δημιουργούμε κοινότητες που κινητοποιούν εμπειρογνωμοσύνη. Το βλέπετε και εδώ. Δύο πλεονεκτήματα από αυτό το μοντέλο. Ε, αντί για 55 ε, έχουμε πλέον ε, μια μόχλευση και έχουμε για να δουλεύουμε για μας πάνω από 300 άτομα. Ε, ταυτόχρονα όμως δημιουργούμε και την ε, αίσθηση ε, της συμμετοχής και σε πάρα πολλούς ανθρώπους εκτός της ενίσα. Αυτό σημαίνει ότι ευκολύνεται η εφαρμογή των συστάσεών μας. Τι κάνουμε. Κάνουμε συστάσεις, εκδίδουμε συστάσεις Εντάξει, χαρτιά βέβαια, κάποιο πρέπει να τα διαβάσει και να τα καταλάβει και αφού τα καταλάβει κάποιο πρέπει να τα εφαρμόσει. Οπότε οι συστάσει είναι μακριά από την πραγματικότητα, το αναγνωρίζουμε, οπότε δεν περιοριζόμαστε στι συστάσει, εργαζόμαστε και στην εφαρμογή πολιτική. Και μάλιστα με τρόπο που θα είναι οικονομικά αποδοτικός. Ε, τι άλλο κάνουμε κάνουμε πρακτική δουλειά, hands-on όπως τη λέμε εμείς, ε, στον τομέα των ε, κυβερνογυμνασίων, κυβερνοδοκιμών. Ε, λειτουργούμε με κοινότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε σε πραγματική, πραγματικό χρόνο να κάνουμε ασκήσεις κυβερνοχώρου και ασκήσεις αντίδρασης. Αυτά είναι τα τρία βασικά συστατικά της δράσης μας. Τρεις διαφορετικοί τύποι δράσεων της ΕΝΙΣΑ. Τώρα, γιατί μιλάμε, σήμερα. Εδώ είμαστε. Ας ξεκινήσουμε τα, με ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα μας ε, που είναι το πανόραμα των απειλών της ΕΝΙΣΑ, οι δέκα μεγαλύτερες απειλές. Ε, δεν ανακοινώνουμε ε, τίποτα εμεί, οι ίδιοι, δεν κάνουμε τίποτα εμεί, οι ίδιοι, παίρνουμε τι έχουν ανακοινώσει οι υπόλοιποι σε όλο τον κόσμο ε, και συνδυάζουμε αυτές τις πληροφορίες ε, έτσι ώστε να τις ταξινομήσουμε, να ταξινομήσουμε τις απειλές ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. Και βέβαια κάνουμε και προβολή αυτών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας μιλούμε για τις κρίσιμες υποδομές πολύ συχνά. Ε, μιλάμε για ε, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ε, συστήματα εφή δίκτυα, οικονομικά, σε υπηρεσίες, που, ε, προσφέρουν οικονομικές υπηρεσίες, πρακτορία, δεσιογραφικά πρακτορία, Reuters κλπ. που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία σε καθημερινό επίπεδο. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό και από την άλλη πλευρά. Οι τράπεζες ενδιαφέρονται πολύ για την ακυρεότητα των δεδομένων τους. Ε, και εγώ από τράπεζα ήρθα. Καταλαβαίνω, αν δεν εξασφαλίσουμε την ακυρεότητα των δεδομένων μας, χάνουμε λεφτά εκεί. Ε, αν όμως βρισκόμαστε σε ένα άλλο κόσμο, στον κόσμο της ε, ε βιομηχανίας, εκεί χρειαζόμαστε συνεχή ε, δυνατότητα πρόσβαση στα δίκτυα ενέργειας για παράδειγμα. Ε, είναι τελείως, διαφορετική, τελείως διαφορετικές οι απειλές εκεί, τελείως διαφορετική η τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις απειλές. Είναι πολύ σημαντικό ε, επίσης να φέρνουμε απομακρυσμένα μεταξύ τους κράτη μαζί έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν από κοινού τις απειλές. Οπότε ε, θα δείτε τελείως ε, ε, διαφορετικό λεξιλόγιο να χρησιμοποιείτε ανάλογα με το σε ποιον μιλάμε. Εδώ και πολλά χρόνια μιλάμε με τα κράτη-μέλη για θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η Εστονία ήταν η πρώτη από το 2008, τώρα πια όμως ε, ε, ε, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν εθνικές στρατηγικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Το λέω αυτό με περηφάνεια. Αυτές οι στρατηγικές ε, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δείχνουν ότι τα κράτη-μέλη προφανώς έχουν διαφορετικό, διαφορετική οριμότητα ε, λογικό. Ε, η στρατηγική ασφάλεια των βασικών υποδομών όμω είναι βασικό σημείο σε όλες αυτές τις ε, στρατηγικέ. Η συνεργασία ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα είναι περιορισμένη αλλά δουλεύουν πάνω σε αυτήν. Θα πρέπει να δούμε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτή η συνεργασία στο μέλλον. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο σκελετός της ε, οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξακολουθούμε να τη στηρίξουμε και βλέπουμε και άλλα θέματα στις στρατηγικές αυτές. Είναι δύσκολη η διακυβέρνηση αυτών των πολιτικών, για παράδειγμα, των στρατηγικών, συγγνώμη, αλλά τούτου λεχθέντος είναι κάτι που οριμάζει στην Ευρώπη, έχει ήδη οριμάσει και θα πρέπει να το προχωρήσουμε. Οι εθνικές στρατηγικές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τώρα, ε, εδώ αναμειγνύω συστήματα κρίσιμων πληροφοριών με την ανταλλαγή και το διαμεσμό πληροφοριών. Ε, είναι κάτι που λαμβάνει χώρα σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ε, οι κοινοποιήσεις περί παραβίασης των μέτρων ασφαλείας, security breach όπως λέμε. Ε, αυτό έχει γίνει, οι τέτοιου κοινοποίηση είναι πλέον υποχρεωτικό στις ΗΠΑ και ε, ετοιμαζόμαστε και στην Ευρώπη ε, με την οδηγία NIS. Κάποιοι πίστευαν ότι θα είναι πολύ κοστοβόρο, δαπανηρό, Πλην όμως ε, στην ε, πράξη αποδεικνύεται ότι ε, εκεί που έχει εφαρμοστεί συμφαρμόζεται πολύ μικρό κόστος για παράδειγμα στις, στις εταιρείε τηλεπικοινωνιών και ταυτόχρονα παίρνουμε και πάρα πολλές πληροφορίες από τις κοινοποίησεις αυτές. Όταν πρωτομίλησα με τους με επαγγελματίες της ασφάλειας για τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε ξεπλάγησαν. Και πάλι όμως αυτοί οι εμπειρογνώμονες δεν θα μπορούσαν να απαντήσουν ποιο είναι ο, ποιος είναι ο νούμερο ένα κίνδυνο για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Ε, κάποιοι νομίζουν ότι είναι κυβερνοεπιθέσει κλπ. Όχι, καμία σχέση τελικά, <laughs> αν δούμε τα αποτελέσματα. Ε, εδώ φαίνεται από πού, είναι τα προβλήματα, πού προέρχονται τα προβλήματα. Και είναι στοιχεία που έχουν προκύψει από αυτέ τι ανακοινώσει παραβίαση των ε, κανόνων ασφαλεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα, οι κόκκινε στήλε είναι απώλειες συστήματος ε, που έχουν προκύψει από hardware ή από software. Εκεί, αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή, ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν το software μας ήταν καλύτερο, θα μπορούσαμε να ε, ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο, η δεύτερη απειλή, το μπλε, είναι ο κακόβλος κώδικας ή οι κυβερνοαπειλές. Δεν λέω ότι αυτός είναι μικρός κίνδυνος, απλά πρέπει να το δούμε σε σύγκριση με κάποιον άλλον που είναι ακόμα μεγαλύτερος επί Ε, υπάρχουν και οι κοινοποιήσεις ε, ε, ε πρόσβασης σε δεδομένα ε, που είναι κάτι διαφορετικό. Ε, αν δηλαδή μια εταιρεία διατηρεί στοιχεία άλλων έχει και την υποχρέωση να ενημερώσει αυτούς τους ανθρώπους αν αυτά τα στοιχεία έχουν κλαπεί ή κάποιο έχει αποκτήσει παρανόμω πρόσβαση σε αυτά. Είναι πολύ σημαντικέ και αυτέ οι κοινοποιήσει και αποτελούν ε, κομμάτι και της ε, οδηγίες περί ε, απορρίτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, στο νέφος. Και εδώ, για το υπολογιστικό νέφος, έχουμε κάνει δουλειά. Ξεκίνησαμε το 2009 με την Cloud Security Alliance με ένα μοντέλ, με ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει τη σύγκριση με βάση συγκεκριμένους, συγκεκριμένες παραμέτρους. Ε, τα προβλήματα στο υπολογιστικό νέφος έχουν και πάλι σχέση πιο πολύ με τις διαδικασίες. Ξέρεις ποιος έχει την ευθύνη της τάδε λειτουργίας, ε, πού τηρούνται τα ε, δεδομένα, είναι στην Κίνα μήπως τα δεδομένα στο νέφος και τι γίνεται εκεί, κάνουμε κανόνες από ό,τι εδώ. Μιλάμε για προβλήματα που προκύπτουν δηλαδή από τη λειτουργία του νέφους. Είναι σημαντικό όμως να καταλάβουμε ε, την σχετική σημασία του κάθε προβλήματος έτσι ώστε να μπορούμε να προστατευτούμε ανάλογα. Εδώ ε, σκάντα είναι τα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, ε, παροχής ενέργειας, ε, χημικές βιομηχανίες κλπ. Έχουμε δουλέψει εδώ και 3-4 χρόνια στο θέμα της προστασία των συστημάτων τους. Εκεί αυτά τα συστήματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα συνεχώς, το οποίο σημαίνει ότι πολύ συχνά αυτοί λειτουργούν με παλιά συστήματα που είναι σταθερά μεν γιατί έχουν αποδείξει την χρησιμότητά τους πολλά χρόνια χρόνια. Από την άλλη μεριά όμω είναι λίγο πεπαλαιωμένα και έχουν μεγαλύτερου ε, κινδύνους, ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους και τις κυβερνοεπιθέσεις. Είναι όμως πολύ σταθερά συστήματα γιατί λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ε, το οποίο σημαίνει ότι βοηθούν τους διαχειριστές να εξασφαλίσουν συνεχή παρουσία και λειτουργία τους. Τώρα, το βασικό μας project είναι οι ασκήσεις κυβερνοασφάλειας. Ε, μας το ζήτησε η Κομισιόν με, μια ανακοινωσή της το 2009. Και ενέπνευσε τα κράτη-μέλη. Από την αρχή ήταν πάρα πολύ δημοφιλέ το πρόγραμμα αυτό. Κάνουμε πραγματικέ ασκήσει γυμνάσια δηλαδή. Αν ήμασταν σε στρατιωτικό περιβάλλον, θα λέγαμε γυμνάσια. Ε, με συγκεκριμένο με συγκεκριμένα σενάρια τα οποία δεν γνωρίζουν οι συμμετέχοντες για να διαπιστώσουμε ε, πόσο ασφαλή είναι τα συστήματά μας. Η πρώτη έγινε το 2011. Ε, συμμετείχα τότε και στην ομάδα. Ε, αποφάσισαμε να ε, δοκιμάσουμε, εξετάσουμε τρία πράγματα. Σε περίπτωση κυβερνό απειλής. Για παράδειγμα, από την Πορτογαλία στις Βρυξέλλες. Μια επίθεση. Ε, δεύτερο, Ε, ε, πώς ξέρετε με ποιον θα πρέπει να μιλήσετε σε τέτοιου είδους περίπτωση. Τρίτον, πώς ανταλλάσσετε πληροφορίες, με ποια κανάλια και πώς μπορούν αυτές οι πληροφορίες να είναι ασφαλείς. Και στα τρία ήταν άσχημα τα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά ήταν καλό, διότι καλύτερα να αποτύχουμε σε μια δοκιμή, σε μια άσκηση, παρά στην πραγματική ζωή. Από, τότε έχουμε κάνει και άλλες ασκήσεις. Θα κάνουμε και μία άσκηση φέτος, ε, πολύ πιο περιπλοκή, ίσως τη μεγαλύτερη στον κόσμο. Όλα τα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν με παρατηρητές. Ε, είναι ένας κύκλος δύο ετών προγραμματισμού, ε, ο οποίος θα ακολουθεί από μια άσκηση με τρεις φάσεις, και τακτική και στρατηγική φάση. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη μας μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και με, τις, ε, με την εμπειρία μας βοηθούν αυτούς που σχεδιάζουν πολιτική. Προκειμένου να βελτιώσουμε την αντίδρασή μας σε τέτοιου είδους κυβερνοεπιθέσεις, βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία, στοιχεία πραγματικού χρόνου, σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες. Και περνάω στο τελευταίο θέμα, η οδηγία NIS, ε, ασφάλειας ε, δικτύων και πληροφοριών. Ε, προέρχεται από τον πυλώνα 1 της ε, στρατηγικής κυβερνοασφάλειας ε, ε, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που δεν σημαίνει τίποτα βέβαια από μόνο του. Κάτι θα πρέπει να, από κάτι θα πρέπει να ακολουθείτε στην πράξη και στην εφαρμογή της οδηγίας ΕΝΑΕΣ κρύβεται ε, το, η ουσία και εκεί η Ενίσσα θέλει να βοηθήσει έτσι ώστε η θεωρία να γίνει πράξη τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να υιοθετήσουν εθνική στρατηγική ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, ε, υποχρεώνονται να ορίσουν τα κράτη-μέλη ε, αρμόδιες αρχές και ομάδες αταχές αντίδρασης, δημιουργεί την πρώτη, ε, το πρώτη, ομάδα συνεργασίας Ευρωπαϊκής για την ασφάλεια δικτύων και ε, πληροφοριών και καθορίσει συγκεκριμένε απαιτήσει ό,τι αφορά τις ε, κοινοποιήσει και την ασφάλεια των ε, διαχειριστών ε, συστημάτων κρίσιμων υπηρεσιών και παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών. Εδώ έχουμε δεξιά τις υπηρεσίες, τις κρίσιμες υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμοδίες των κρατών μελών, καταλαβαίνετε μεταφορές, ενέργεια, ίδρυυση, υγεία κλπ. Τώρα και μπορούμε να βοηθήσουμε και, και εκεί, αν μας ε, ζητηθεί, γι' αυτό είμαστε και εμείς δεξιά. Αριστερά είναι αυτά για τα οποία έχουμε εφαρμοστικές πράξεις και βοηθούμε την Κομισιόν να εφαρμόσουν τις τα αντίστοιχα άρθρα της οδηγίας. Ε, οπότε, παρόλο που δεν έχει υιοθετηθεί, έχει, έχει συμφωνηθεί, οπότε εμείς είμαστε ήδη δραστήριοι, έτσι ώστε να είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη να τη μεταγράψουν όταν χρειαστεί. Τελειώνω με ένα ακόμα στοιχείο. Ε, υπάρχει ιδέα, μάλλον ε, η δυνατότητα η ΕΝΙΣΑ να, ε, να υποστήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην δημιουργία κρίσιμων ε, υποδομών. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μην πέστε στην παγίδα να πιστεύετε ότι η ανταλλαγή περισσότερων πληροφοριών είναι καλύτερη, είναι πιο ωφέλιμη. Όχι απαραίτητα εξαρτάται ποιε είναι αυτέ τι πληροφορίε. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μόλυνση δεδο, με δεδομένα, πάρα πολλά δεδομένα, υπερπροσφορά. Ε, οπότε το τρίκ στο μέλλον, το κόλπο είναι στο μέλλον, οι πληροφορίε να ανταλλάσσονται με το σωστό τρόπο, τη σωστή στιγμή, σωστέ πληροφορίε για να πάρουμε τα σωστά αποτελέσματα. Αλλά πρώτα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα σωστά αποτελέσματα και μετά να πάμε προ τα πίσω. Προφανέ, αυτονόητο δείχνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, πολλέ φορέ κάνουμε λάθο. Συμπεράσματα συνεργαζόμαστε με κοινότητες, επιχειρησιακές κοινότητες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εντοπίζουμε τις ε, ρεαλιστικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα ασφάλειας. Ε, εκδίδουμε συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια και ποιες εφαρμογές να, πρέπει να προτιμηθούν. Οι, προ... η προτείνουμε βασίζονται στις καλύτερες, στις βέλτιστες πρακτικές και δουλεύοντας με αυτόν τον τρόπο βάζουμε την ασφάλεια την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας και της οικονομίας μας γενικά. Η, συνεργασία μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού πολιτικού τομέα ε, θα γίνεται όλο και πιο σημαντική στο μέλλον και θα πρέπει ο ένας να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα του άλλου προκειμένου να εξασφαλίσουμε οριζοντίως την ασφάλεια σε όλες τις χώρες και σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σα. Ε, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ορισμένε από τι δηλώσεις ε, εδώ για τη ΣΕΝΤΕ, ειδικότερα οι τρόποι ε, κοινοποίησης των πληροφοριών. Να σας ακούσουμε τώρα και την άποψη του ΝΑΤΟ, ο κύριο Κρίστιαν Μαρκ Λιφλέντερ από το ΝΑΤΟ. Έχει το λόγο αυτή τη στιγμή. Καλημέρα. Να ξεκινήσω κι εγώ με τις ευχαριστίες μου που με καλέσατε να συμμετέχω σήμερα εδώ και ευχαριστώ που ενδιαφερθήκατε για την άποψη του ΝΑΤΟ. Ε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, ε, ο κυβερνοχώρος ε, δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνολογίας, αλλά είναι και ζήτημα πολιτικής. Ξεκινώντας την ομιλία μου θα σας αναφέρω δύο παραθέσεις. Η πρώτη προέρχεται από την Sony Pictures Entertainment και τον πρόεδρό της. Είπε ότι στο διαδίκτυο ε, δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Ουσιαστικά κοιτάει την κατάσταση κανείς. Απλά και μιλούσε για την επίθεση ε, μέσω διαδικτύου στα Sony Studios Κοιτάει λοιπόν κανείς την κατάσταση και δεν έχει και μεγάλη εμπειρία για να χρησιμοποιήσει. Ε, απλά χρησιμοποιεί ό,τι υπάρχει από εμπειρία. Η δεύτερη παράθεση είναι από τον Eric Schmidt, ε, τον πρόεδρο της Google. Είπε λοιπόν ότι το διαδίκτυο είναι το πρώτο πράγμα που έχτισε η ανθρωπότητα, αλλά το οποίο δεν καταλαβαίνει το μεγαλύτερο πείραμα που κάναμε ποτέ. Αυτές οι δύο παραθέσεις πιστεύω συνοψίζουν πολύ σωστά τη φύση και την τρέχουσα κατάσταση του διαδικτύου. Ε, η διασύνδεση ε, στον κυβερνοχώρο φυσικά προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την παγκόσμια οικονομία και μετασχηματίζει τη φύση των κοινωνιών μας, αλλά χαρακτηρίζεται και από κάποιο βαθμό χάους. Αυτός ο διασυνδεδεμένος χώρος μας καθιστά ευάλωτους καθώς αυξάνεται η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο δυσκολεύοντας την ασφάλεια όλο και περισσότερων μηχανημάτων. Για να είμαι πιο ακριβής, οι επιθέσεις είναι ταχύτερες από ότι εμείς οικοδομούμε την αμυνά μας. Σκόπιμο είναι λοιπόν να σταματήσουμε να συζητάμε άμυνα στον κυβερνοχώρο σαν να υπερασπιζόμαστε ένα κάστρο χτίζοντας ένα τείχο γύρω του. Όπως τα πράγματα έχουν τώρα, η ανείχνευση είναι αυτή που έχει αντικαταστήσει την άμυνα ως στρατηγική, ώστε έτσι λοιπόν για να είμαστε αποτελεσματικοί, η άμυνα πρέπει να είναι ανθεκτική και αρκετά ευρηματική, ώστε να μπορεί να αμυνθεί, να προστατεύσει ένα σύστημα, να περιορίσει τις επιπτώσεις και να βοηθήσει στην ε, ανάκτηση της λειτουργικότητας των ταχύτερων δυνατών. Όσον αφορά τον κυβερνοχώρο, θα το έχετε ακούσει ήδη, το ακούσετε ήδη από τον Ενίσα και ε, από τον Στίβ. Ξέρετε, υπάρχουν τόσο πολλοί κακόβουλοι ε, ε, άνθρωποι ε, στο κυβερνοχώρο, έχουμε οργανωμένο έγκλημα, ακτιβιστές, ε, αλλά και κυβερνήσεις, ανθρώπους ε, ε, που, ανθρώπους που χορηγούνται από κράτη για, κακόβουλες, για κακόβουλους σκοπούς. Οι τεχνικές, έχουμε το spear phishing και web compromises, τα οποία είναι τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των χρηστών με την κλοπή του ονόματος χρήστη του κωδικού πρόσβασης ή με την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού υπάρχει ε, η ε, χειραγώγηση χρηστών ε, για την πραγματοποίηση δράσεων που παρέχουν τα στοιχεία κάποιου χρήστη, σε κάποιον κοβλού χρήστη. Επίσης υπάρχουν λογισμικά ιδιαίτερα σχεδιασμένα για καταστροφή υπολογιστικών συστημάτων ή worms και τα trojans τα οποία βρίσκονται σε διαρκή αύξηση. Και θα είδα τα στατικά στοιχεία της ΕΝΗΣΑ. Ε, πολύ καλή ήταν η παρουσίασή σας, μάλιστα ήταν πολύ επιτυχηματική. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο είναι προηγμένη τεχνολογίες επιθέσει ε, και επίμονες επιθέσει που απαιτούν τεράστια χρηματοδότηση, τεχνική προγνωμοσύνη και εξειδικευμένε γνώσει ε, του στόχου αυτέ. οι δραστηριότητε, οι οι προηγμένε έμόνε απειλέ. Ε, στοχεύουν συχνά κράτη, υπουργεία εξωτερικών, πρεσβείες, ε, ε, κοινοβούλια κτλ. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, εμείς ασχολούμαστε με την ασφάλεια εδώ και 67 χρόνια. Η δυναμή του άρθρου 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, η επίθεση προς ένα μέλος είναι επίθεση προς όλους. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη υπόσχεση ότι τα κυρίαρχα κράτη μπορούν να βοηθήσουν το ένα το άλλο. Δεν είναι απλά κάτι γραμμένο σε χαρτί. Έχουμε χτίσει έναν τεράστιο διεθνή οργανισμό ώστε να μπορέσουμε να καταστήσουμε πιστευτή αυτή την υπόσχεση. Ε, μιλάμε για έναν οργανισμό με μία μόνιμη διαδικασία πολιτικής διαβούλευσης και έναν εξελιγμένο ε, μηχανισμό απόκρισης και δίκησης. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να παρέχει κανείς ε, αξιόπιστη ασφάλεια Το ΝΑΤΟ έχει στις προσδοκίες, είτε προκτώ για την αποτροπή κατά τον ψυχρό πόλεμο της Σοβιετικής Ένωσης, να τερματίσει τον πόλεμο ε, στο ε, Βαλκάνια, αλλά παρά αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα χρειάστηκε μία απότομη αφύπνιση για να εστιαστούμε στις, ε, στα θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου και όπως αναφέρθηκε αυτή η αφύπνιση προήλθε από τις επιθέσεις στην Εστονία του 2007. Τι συνέβη στην Εστονία. Η Εστονία για τον ΝΑΤΟ και όλα αυτά που συνέβησαν εκεί ήταν κάτι νέο. Για πολλά χρόνια είχαμε εστιαστεί στην άμενα. Δηλαδή ουσιαστικά βγάζει όπλα κανείς απλά για να δείξει ότι έχει τη δύναμη χωρίς να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά είδαμε ότι στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αυτό δεν αρκεί. Έπρεπε να προσθέσουμε σε αυτό την πτυχή της, ασφ... πρόληψης και ακόμη περισσότερο σημαντικό της αντοχής. Με άλλα λόγια, αν δεν μπορούμε να προλάβουμε την κάθε επίθεση, πρέπει να προσπαθήσουμε να παρεμποδίσουμε τον επιτιθέμενο από το να αποκτήσει οποιοδήποτε κέρδος και να ανακτήσουμε τις λειτουργίες μας το ταχύτερο δυνατόν. Μια τέτοια στρατηγική περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία όσον αφορά μας τον ΝΑΤΟ. Πρώτον, τις ικανότητες. με την έγκριση τη ενισχυμένη πολιτική του ΝΑΤΟ για την άμυνα στον κυβερνοχώρο στην, ε, στο συνεδρίο μα στην Ουαλία πριν δύο χρόνια αναγνωρίστηκε ότι η αρχή τη συλλογική άμυνα αφορά επίση και τι απλέ του κυβερνοχώρου. Ουσιαστικά αυτό αφορά το άρθρο 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου που αποτελεί το βασικό θεμέλιο του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι όπω εμεί καταλαβαίνουμε τον κυβερνοχώρο αυτό αποτελεί μια μεγάλη εξέλιξη. Αναφέρθηκε πρώτη φορά το 2010 στη στρατηγική μας ε, ε, ε, θεωρία ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να απειλήσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον χώρο του Βορειοατλαντικού. Το θέμα είναι ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο σοβαρές για τις κοινωνίε μας όσο και οι κλασικέ ε, στρατιωτικέ επιθέσεις. Έτσι λοιπόν η άμυνα στον κυβερνοχώρο έχει αναγνωριστεί ρητά ως κομμάτι της συλλογική άμυνας του ΝΑΤΟ. Ίσης σημασίας. Ε, αυτό ε, επικοινωνείται από το γεγονό ότι και το διεθνέ δίκαιο εφαρμόζεται στον κυβερνοχώρο. χώρο ε, μην ξεχνά τα θέματα διαφάνειας ε, και κριτικής ενίσχυσης. Για μας λοιπόν δεν είναι πλέον άγνωστο έδαφος, ε, δεν είναι far west αυτό, αυτός ο χώρος και ειδικότερα όσον αφορά τη χρήση δύναμης κτλ. Πώς αποφασίζουμε πότε ενεργοποιείται το άρθρο 5 σε περίπτωση μιας επίθεσης στον κυβερνοχώρο, αυτό απαιτεί πολιτική απόφαση που θα ληφθεί από το ΝΑΤΟ κατά περίπτωση. Το γνωρίζουμε δηλαδή με άλλα λόγια μόλις το δούμε. Και είναι μια κρίση πολιτική, πολιτικού χαρακτήρα. Για να είμαστε σίγουροι ότι το ΝΑΤΟ θα μπορέσει να εκπληρώσει αυτό το βασικό καθήκον της άμυνας στον κυβερνοχώρο, χρειαζόμαστε τις απαραίτητες δυνατότητες και ικανότητες τόσο εντός του ΝΑΤΟ όσο και σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν για το ΝΑΤΟ υπήρξε προστασία των δικών του δικτύων. Ακούγεται εύκολο, αλλά δύσκολο στην εφαρμογή, αλλά ξέρετε το ΝΑΤΟ είναι ένας ιδιαίτερος διεθνής οργανισμός, γιατί έχει τα δικά του δίκτυα σε ολόκληρη ε, τη γη, από τη Νορβηγία μέχρι τη Μεσόγειο και από τη Βόρεια Αμερική μέχρι το Αφγανιστάν. Δεν είναι και κάτι εύκολο να προσθέσω. Με άλλα λόγια, το ΝΑΤΟ εστιάζεται σε αυτά τα δίκτυα και στην προστασία τους. Ενώ οι σύμμαχοι ε, προσπίζουν τα δικά τους. Και το βασικό μας εργαλείο είναι το, μέσο που, το εργαλείο που έχουμε για την προστασία των δικών μας συστημάτων. Όσον αφορά την άμυνα των συμμαχών, εμείς ε, δρούμε ως διαμεσολαβητές. Ο σχετικός μηχανισμός είναι η διαδικασία σχεδιασμού άμυνας του ΝΑΤΟ. Επίσης, ε, η κοινή χρήση πληροφοριών είναι ένα σημαντικός παράγοντας μεταξύ των συμμάχων και με εμάς. Και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα των εργασιών μας, με στόχο να βελτιώσουμε την πρόληψη και την αντοχή κατά απειλών στον κυβερνό χώρο, ε, δίνοντας περισσότερη σημασία σε αυτές τις εργασίες. Για να οικοδομήσουμε ικανότητε. εστιαζόμαστε στην εκπαίδευση, στι ασκήσεις και στην κατάρτιση. Για παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων ε, ε, για άμυνα στον κυβερνοχώρο. Αυτό συνεπάγεται εκπαίδευση προσωπικού ε, σε διαδικασίες αλλά και τεχνολογία. Οπότε εμείς θέλουμε να εστιαστούμε στην πρόληψη και στην αντοχή στην πηγή. Ο δεύτερος πυλώνας, ίσως πιο σημαντικός, είναι ευρείες συνεργασίες. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι ο κυβερνοχώρος είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ότι η άμυνα στον κυβερνοχώρο είναι μια συνεργατική προσπάθεια. Οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών είναι τομεί στου οποίου αφορά η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ένα μεγάλο κομμάτι του κυβερνοχώρου βρίσκεται εκτό του ελέγχου των κυβερνήσεων. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με μια τεράστια ε, παγκόσμια συμμαχία που υπερβαίνει τις κυβερνήσεις ε, και περιλαμβάνει και ε, τα πανεπιστήμια και τους διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Όσον αφορά τους βιομηχανικούς τομείς, τον τομέα των υπολογιστών, να γνωρίζουμε ότι η βιομηχανία είναι ένας βασικός παίκτη στον κυβερνοχώρο. Είναι κάτοχοι των μεγαλύτερων υπολογιστικών συστημάτων του κόσμου, αλλά παρέχουν και τεχνικές λύσεις για την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Γιατί, διότι ένα μεγάλο κομμάτι της καινοτομίας ε, προέρχεται από τη βιομηχανία και βασίζεται στις δικές της τεχνολογίες και τη δική τους εμπειρογνωμοσύνη. Γι' αυτό η εταιρική σχέση με αυτούς είναι αναγκαία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο διαδικασία. Ε, είναι αρκετά δύσκολο, είναι πολύ πιο δύσκολο στην πρακτική παρά στα λόγια, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης αποτελεί προτεραιότητα για μας. Όπως ε, επισημάνθηκε νωρίτερα εδώ από τη Χέλη, έχουμε συνομιλίες μεταξύ των αντίστοιχων επιτροπών για να μοιραζόμαστε πληροφορίες και να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, λέει η κυρία Πρόεδρος. Και προβαίνουμε σε συνέργειες όποτε αυτό είναι δυνατόν. Ουσιαστικά πρακτικά αυτό που φτιάξαμε το Φεβρουάριο είναι μια τεχνική συμφωνία που θα μας επιτρέψει με πιο πρακτικό τρόπο να προλαμβάνουμε τις επιθέσεις στον κυβερνό χώρο αλλά και να βελτιώσουμε τη δυνατότητα πρόβλεψης, ανείχνευσης και απόκρισης της επιθέσεις στον κυβερνό χώρο. Ένας όλος τρόπος ε, που ανέφεραν και οι προλαλήσαντες είναι να ενισχύσουμε ε, τη δυνατότητα κοινών ασκήσεων άμυνα στο κυβερνοχώρο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κληθεί να παρακολουθήσει τις ασκήσεις του ΝΑΤΟ ε, στο πρόγραμμα μας Cyber Collision και παρομοίως στο ΝΑΤΟ. Μόλις ετοιμαστεί το Cyber Europe φαντάζομαι Ενδεχομένω θα κληθεί να συμμετάσχει στη σχετική άσκηση. Τώρα για να κλείσουμε από αυτή τη σύντομη παρουσίαση παρατηρούμε ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά. Αντιλαμβανόμαστε το επίγον του ζητήματος και δρούμε ανάλογα τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή κατά την απόψή μου μίας μάλλον μακροχρόνιας ε, ε, δύσκολη και ενδιαφέρουσα διαδικασία. Όπω είπα στην αρχή τη παρουσίασή μου, η άμυνα στον κυβερνοχώρο είναι λίγο χαόδη. Διότι δεν αντιστοιχεί στα κλασικά μοτίβα απειλή και ανταπόκριση ε, στρατιωτική φύση που είχαμε, ούτε στα μοτίβα που είχαμε για την εσωτερική ασφάλεια ενό κράτου. Με στου επόμενου μήνε, καθώ προετοιμαζόμαστε για τη Σύνοδο Κορυφή ε, του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, οι σύμμαχοί μας θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται στις νέες πραγματικότητες και δεδομένου του δυναμικού διεθνούς περιβάλλοντος. Το ΝΑΤΟ είναι σημαντικό για την συλλογική μας ασφάλεια περισσότερο από ποτέ. Πιο συγκεκριμένα υλοποιούμε το σχέδιο ετοιμότητας ε, για καταστάσεις επίγουσας ανάγκης ως απόκριση για την επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τριπλασιάζουμε τη δύναμη απόκρισης του ΝΑΤΟ σε 30.000 άτομα που μπορούν να αναπτυχθούν εντός 24 ώρων, εντός 48 ώρων. Παρομοίως, στη μη στρατιωτική πλευρά, η άμυνα στον κυβερνοχώρο θα συμπεριλαμβάνεται διαρκώς στην ατζέντα του ΝΑΤΟ. Για να το πω απλά, είναι αδύνατο να φανταστώ μια μελλοντική διαμάχη που δεν θα έχει και μια συνιστόσα στον κυβερνοχώρο. Σε αυτό το περιβάλλον λειτουργούμε σήμερα, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και σήμερα και στο μέλλον. Αυτά ήταν η ομιλία μου. Σας ευχαριστώ και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Πρόεδρο. ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την ε, τόσο πλήρη και σαφή παρουσίαση. Τώρα, συζήτηση. Ο κύριος ε, Τουνεκέλεμεν ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις εξαιρετικές σας παρουσιάσεις. Όπως είπε και ο κύριος Λίφλαντερ, εξακολουθεί να είναι αχαρτογράφητα νερά για μας. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα καταρχήν. Έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τη συνεργασία, μετά με την οικοδόμηση ικανοτήτων και τρίτον με τα μέσα που διαθέτουμε για την οικοδόμηση αυτή ικανοτήτων αναφερθήκατε στη δημιουργία ενός δικτύου επαφών. Αναρωτιέμαι λοιπόν, όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, έχουμε παντού συμπεριλάβει και την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Στις συμφωνίες δηλαδή που κάνουμε με τρίτες χώρες συμπεριλαμβάνεται. Έπειτα, για την εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού. Ποια είναι τα κύρια εμπόδια που παραμένουν. Η τι εξελίξεις έχουμε. Αναφερθήκατε στη συνεργασία για το υπολογιστικό νέφος. Είναι ένα θετικό βέβαια παράδειγμα. Υπάρχουν άλλα τέτοια παραδείγματα συνεργασίας. Και κάτι ανησυχητικό. Είναι το θέμα των στρατηγικών, των εθνικών στρατηγικών για την ε, κυρνευοασφάλεια. Το ότι δηλαδή είναι σε τελώς διαφορετικό βαθμό προετοιμασμένες οι χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν απειλές στον κυβερνοχώρο. Και το πιο βασικό είναι η έλλειψη πόρων ή όπως αναφερθήκατε κι εσείς η ενίσα πιο συγκεκριμένα ότι ο προπολογισμό σας είναι ψίχουλα. Άννα, μιλάμε σοβαρά για τις απειλές αυτές, πόσο σοβαρές είναι οι ίδιες, πόσο μεγάλες είναι οι απειλές, δεν είναι δυνατόν να μένουμε στη διαμαρτυρία. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι οι πόροι δεν ανταποκρίνονται στο μέγεθος των αναγκών. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να στηρίξουν την κατάλληλη χρηματοδότηση για να οικοδομήσουμε τις ικανότητές μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Έργαν Φλόιντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που άργησα να φτάσω στη συνάντηση. Σίγουρα ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις πριν φτάσω. Θέλω όμως να αρχίσω με μία παράθεση που λέει το εξή. Φανταστείτε ένα blackout που κρατάει εβδομάδες και μήνες. Ε, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο που δεν έχουν πρόσβαση σε γεννήτρια και υπάρχουν ε, πολλές τέτοιες περιπτώσεις που δεν έχουν ε, νερό, φάρμακα τράπεζες δεν θα λειτουργούν πια και η δημόσια τάξη δοκιμάζεται όπως ποτέ στο παρελθόν. Δεν πρόκειται απλώς για ένα σενάριο. Είναι μια καλά σχεδιασμένη επίθεση στα διάφορα δίκτυα ενέργειας που θα πλήξει όλους μας τις υποδομές. Και στην εποχή του ηλεκτρονικού πολέμου καταλαβαίνετε ότι μόνο αν έχουμε τα μέσα να τον αντιμετωπίσουμε ε, μπορούμε να προστατευτούμε. Είναι μια παράθεση. Ο Τετ που είναι φίλος μου και είναι δημοσιογράφος Αμερικανός και παρουσιαστής ε, παλιότερα στην τηλεόραση, πριν από ένα χρόνο έγραψε ένα βιβλίο που έλεγε «Έσβησαν τα φώτα». Όπως καταλαβαίνετε, αφορά ακριβώς τέτοιου είδους σενάρια ηλεκτρονικού πολέμου, που όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να συμβεί είτε στην Ευρώπη, είτε στις Ηνωμένε Πολιτείε, με την εξαίρεση βέβαια ότι τα δικά μας τα δίκτυα δεν είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα όπως θα θέλαμε από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση αυτού του ηλεκτρονικού πολέμου, γιατί αν επιτεθεί κάποιος στα δίκτυα μιας χώρας, αυτό δεν σημαίνει ότι τα δίκτυα σε ολόκληρη την Ευρώπη υποφέρουν εξίσου. Τότε, από αυτά που συζητήσατε, κατάλαβα λίγο πολύ τι εννοείται. Τώρα, μήπως κάποιος από εσά γνωρίζει να υπάρχει κάποιο σχέδιο για να αντιμετωπιστούν αυτές οι φοβερές προκλήσεις που θα επηρεάσουν ή επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αντίστοιχα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ο επόμενος ομιλητής, κύριος Μαρικίτσερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαρίστως να πάρω κι εγώ το λόγο. Ίσως θα μπορούσα να σας ζητήσω να μας δώσετε τον κατάλογο των απειλών με την σημασία που έχουν. Πρώτα τις πιο σημαντικές και σιγά σιγά τις λιγότερο σημαντικές απειλές που έχουμε στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Έχουμε συνέχεια απειλές. Η διεθνής ε, κρίση όμως απαιτεί να γνωρίζουμε και τι ιδιωτικές πρωτοβουλίες επηρεάζουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η κατασκοπία είναι μία πτυχή αυτού του ζητήματος. Επί το ενεργειακού πολέμου, τα δίκτυα, όπως λέγαμε και πριν. Μπορεί μια τέτοια επίθεση να αποτελέσει μέρος μιας γενικότερης σύγκρουσης. Και αυτό με φέρνει και σε ένα τρίτο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω. Το ρώτησε και ο προλαλής σας. Η απειλή ενδυνάμει απειλή από μια γενικευμένη τρομοκρατική επίθεση. Πώς μπορούν οι τρομοκράτες να επιτεθούν στα δίκτυα ηλεκτρισμού, στα αεροδρομιά μας και τι κλίμακα ζημιά μπορούν να πετύχουν. Βλέπουμε ότι σκοτώνονται άνθρωποι με συμβατικά όπλα, αλλά μπορεί οι τρομοκράτες να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν και άλλες μορφές όπλων. Το έχετε σκεφτεί, πώς βλέπετε εσείς αυτές τις απειλές στο εγγύς μέλλον. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στο πάνελ, θέλω κι εγώ να ρωτήσω κάτι. Και να ρωτήσω και τους τρεις σας, αν μη τι άλλο, την κυρία τίρμα Κλάρ, και τον κύριο Λιφ Λάντερ, να μας πούν σε τι βαθμό μπορεί να εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο, σε περίπτωση συγκρούσεων ασυμμετρικών ε, πολέμων συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού. Γιατί καλά οι κρατικοί παράγοντες, οι μη κρατικοί παράγοντες όμως προφανώς δεν τηρούν το διεθνές δίκαιο. χρησιμοποιούνται τα παιδιά πολλές φορές στην Αφρική. Απαγάγουν τα παιδιά οι τρομοκράτες και τα χρησιμοποιούν στη συνέχεια για να κάνουν επιθέσεις ή επιθέσεις που γίνονται σε νοσοκομεία. Τέτοια είδους προβλήματα, τι δυσκολία προκαλούν στην αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού πολέμου και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα διάφορα μέρη. Πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιες επιθέσεις που γίνονται από ασυμμετρικούς παράγοντες. Λοιπόν, τις απαντήσεις θα αρχίσουμε από την κυρία Κύρμα Κλάρ, με την ίδια σειρά δηλαδή που έγιναν και παρουσιάσεις. Στη συνέχεια ο κύριος Πέρσερ και τέλος ο κύριος Λιφλάντερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολύ καλές σας ερωτήσεις. Ναι, πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να συμπεριλάβει τη διάσταση της ασφαλείας στον κυβερνοχώρο στις ε, ε συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και σε άλλες περιφέρειες και σε άλλες χώρες. Μέχρι στιγμής ε, έχουμε συμπεριλάβει τις παραγράφους για τον κυβερνοχώρο και στο πλαίσιο του διαλόγου με διάφορες ε, χώρες. Ε, και στο διάλογο με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία. Δεν έχουμε κάνει το διάλογο, αλλά έχουμε την παραγραφό στην Συμφωνία Συνεργασία και κατά καιρού ε, συζητάμε το ίδιο με το Μεξικό, την Νότια Αφρική και όλε τι υπόλοιπε οικονομικά σημαντικέ χώρε σε κάθε ήπειρο. Έχουμε περιφερειακέ συμφωνίε με την ΑΣΕΑΝ, με την Μερκοσούρ, με την Αφρικανική Ένωση και με άλλες περιοχές όπου σε αυτές τις συμφωνίες έχει συμπεριληφθεί ο κυβερνοχώρος και σε κάθε νέα συμφωνία φροντίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε μια αναφορά στα ζητήματα του κυβερνοχώρου. Όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία, εκεί προχωράμε και πιο πέρα από μια απλή αναφορά, αναφερόμαστε πιο συγκεκριμένα στην οικοδόμηση ικανοτήτων, την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και σε όλες τις υπόλοιπες έννοιες. Τώρα το κατά πόσο ένα τέτοιο blackout ε, τριών εβδομάδων είναι κάτι ρεαλιστικό. Ξέρετε, έχουμε όλε αυτέ τι ιστορίε τρόμου από του δημοσιογράφου που καλό είναι γιατί ευαισθητοποιούν τον κόσμο, αλλά συζητώντα με του ε, εμπειρογνώμονε που εργάζονται σε τέτοια συστήματα, εάν δεν καταστρέψει πραγματικά κανεί ε, τα μηχανήματα, το οποίο είναι σχεδόν αδύνατον, είναι αμφισβητήσιμο το κατά πόσο θα μπορούσαν να πέσουν ε, οι υπηρεσίε για τρει εβδομάδε συνεχώ. Αν φυσικά κάποιο ιό σβήσει όλα τα δεδομένα, τότε ίσως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποια μη αυτόματα συστήματα. Το πρόβλημα είναι ότι τέτοια συστήματα δεν υπάρχουν πλέον κατά την κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας ε, το Δεκέμβριο τον περασμένο επέστρεψαν στο μη αυτόματο σύστημα διότι υπήρχε ακόμα και είχαν και κόσμο που μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ήξερε πως να το χρησιμοποιήσει και αυτό έζωσε την Ουκρανία ε, την παραμονή των Χριστούγεννων αλλά εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα στα... Έχουμε πολύ πιο προηγμένα συστήματα στη Δυτική Ευρώπη. Οπότε το ερώτημα είναι πολύ ενδιαφέρον και ο Στίβ νομίζω βέβαια από τεχνική άποψη γνωρίζει περισσότερα και μπορούσε, θα μπορούσε να σα απαντήσει αυτό. Ε, για τι τρομοκρατικέ επιθέσει. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι τα πιο επικίνδυνα εργαλεία είναι αυτά που έχουν στην κατοχή τους τα κράτη. Και οι τρομοκράτες δεν χρησιμοποιούν ακόμα εργαλεία καταστροφής, φυσικής καταστροφής των μηχανημάτων μέσω ε, κυβερνοεπιθέσεων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουν να τα αποκτήσουν. Ειδικότερα όταν βλέπουμε τη σύνδεση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ξέρετε, οι επιθέσεις ε, που έγιναν από την ε, από εγκληματικές ομάδες ε, μας απέδειξαν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο ε, όταν έχουμε επιθέσεις που σχετίζονται με ομάδες μαφιόζων. Τώρα το επιχείρημα της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου είναι πολύ καλό το ερώτημα αυτό. Ευχαριστώ που το αναφέρατε. Εμείς αναρωτιόμαστε πώς θα γίνει η εφαρμογή του διεθνούς, ε, ανθρωπιστικού, ε, του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σχετικού χάρτη στον κυβερνοχώρο ήδη από το 2009. Δεν είναι μυστικό ούτε για, ε, ότι έχουμε ξαναεργαστεί στη, με την κυβέρνηση της Εστονίας και υπάρχει το εγχειρίδιο του Ταλίν. Κάτι που ξεκινήσαμε στην Εστονία για να αναλύσουμε το εφαρμογή του Διεθνούς ε, Ανθρωπιστικού Δικαίου και στο εγχειρίδιο ε, αποφασίσαμε ότι εφαρμόζεται και στον κυβερνοχώρο με όλες τις προϋποθέσεις εφαρμογής. Το πρόβλημα είναι ότι το εγχειρίδιο του Ταλίν αναφέρεται μόνο για την εφαρμογή του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε περίπτωση διαμάχης, ενώ η ερώτησή σας αφορούσε τους μη κρατικούς παράγοντες και τι είδους δίκαιο ε, εφαρμόζεται όταν υπάρχει μια διαμάχη χωρίς να έχει κηρυχθεί πόλεμος. Τώρα έχουμε το δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου, αυτή είναι η καλή είδηση που θα βγει φέτος, όπου διεθνείς ε, νομικοί αναλύουν το ίδιο ζήτημα. Ποια νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση τέτοιας σύγκρουσης ε, στον κυβερνοχώρο έχουν δανειστεί πολλά ενδιαφέροντα παραδείγματα από την νομοθεσία για την ανοιχτή θάλασσα και άλλους τομείς ε, ε, σε περίπτωση προβλήματος στον κυβερνοχώρο. Όλα αυτά τα ζητήματα αναλύονται εκεί. Τώρα, όσον αφορά την ποιολητική επιχειρηματολογία, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν κάνουμε συζητήσει για τον κυβερνοχώρο, με του εταιρείς μα συζητάμε το ζήτημα αυτό. Και θέλουμε να έχουμε μια κοινή κατανόηση σε όλα τα κράτη-μέλη ε, ότι το διεθνέ δίκαιο θα ε, ισχύει ε, και στι επιθέσει στον κυβερνοχώρο και μεταξύ άλλων και το δίκαιο για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα, για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, παντού. Αλλά φυσικά υπάρχουν χώρες που λένε ότι αυτό δεν αρκεί και ότι χρειάζεται ένας νέος κώδικας διοντολογία για τον κυβερνοχώρο. Θα ακούσατε ότι η Κίνα, η Ρωσία και κάποιε χώρε της κεντρική Ασίας έχουν δημιουργήσει ένα κώδικα διοντολογία ε, στην οργάνωση ε, συνεργασία τη ΑΝΚΑΙ το 2015. Εμείς δεν συμφωνούμε με τα επιχειρήματα αυτά, διότι θεωρούμε ότι για να υπάρχει ένας τέτοιος ε, κώδικας διοντολογία για τον κυβερνοχώρο και η σχετική νομοθεσία πρέπει να έχει επιληθεί πρώτα απ' όλα το ζήτημα τη απόδοση δικαιοδοσίας, διότι είναι δύσκολο να μπορεί να επαληθεύσει κανείς την προέλευση μιας επίθεσης και να ξέρει ποια δικαιοδοσία θα επιλέξει για να εφαρμοστεί νομοθεσία. Όλες αυτές οι προσπάθειες δημιουργίας ε, ενός κώδικα διοντολογίας και μιας συνθήκης ε, ε, πολέμου στον κυβερνοχώρο έχουν ενδιαφέρουσες συνέπειες στις συζητήσεις και επηρεάζουν αρνητικά και τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό δεν συμφωνούμε με τον κώδικα αυτό της Σανγκάη. Οπότε εφαρμοζούμε την ισχύουσα νομοθεσία. Ευχαριστούμε, κύριε Πέσσερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω τις παρατηρήσεις στη σειρά τους. Κύριε Κέλαμ, πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις ε, σχέσεις ε, δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Σε ευρωπαϊκό πεδίο, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι τέτοιε σχέσει χτίζονται σιγά σιγά από μικρό αριθμό ατόμων αρχικά που συναντώνται ζωντανά ε, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήματα ανάπτυξη τέτοιων σχέσεων. Ίσως σε ευρωπαϊκό πέρα το καλύτερο θα ήταν να, κάνουμε, να χτίσουμε μια ε, δομή ομπρέλα που θα δίνει το πλαίσιο για σχέσεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα στα κράτη-μέλη. Ε, η, με αυτόν τον τρόπο ίσως θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Μετά υπάρχει και το θέμα της ε, ανταλλαγής ε, διαμοιρασμού πληροφοριών στο διαδικτύο online, το οποίο είναι ακόμα πιο περίπλοκο, γιατί όταν κάποιος μιλάει με κάποιον άλλον μέσω τηλεδιάσκεψης, δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από την κάμερα και πρώτα πρέπει να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνη ε, με απευθείας επαφές και μετά να κάνουμε τέτοιου είδους διαμοιρασμό. Η σχέση ιδιωτικού, ιδιωτικού με δημόσιο τομέα, ε, οι εταιρικέ σχέσει μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δεν είναι η μοναδική δυνατότητα. Μπορούμε να έχουμε πιο χαλαρέ σχέσει που να μην είναι εταιρικέ σχέσει, να μην είναι PPP δηλαδή, SDIT. Ε, Τώρα, για το υπολογιστικό νέφος ε, έχουμε πολλά παραδείγματα, έχουμε εργαστεί, συνεργαστεί ε, με, με εταιρείε για, σε project μικρού ε, για την ενεργειακή ασφάλεια, το οποίο δεν ανέφερα πριν. Όλοι χρησιμοποιούμε υπολογιστές με software από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, hardware από την Κίνα. Είναι δύσκολο όλα αυτά να τα βάλει κανείς μαζί και να τα αντιμετωπίσουμε τον ίδιο τρόπο. Ε, επίσης, ε, συνεργαζόμαστε πολύ με τον ΕΤΣΙ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης Τηλεπικοινωνιών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μετατρέπουν πολύ πιο εύκολα από εμά τα δικά τους πρότυπα σε πρότυπα του ISO. Αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα χρονικό, οπότε θα πρέπει να δούμε ε, το, την στρατιωτική προσέγγιση, πώς τα καταφέρνουν και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε πολύ γρήγοροι γιατί έχει σχέση αυτό με το, τα μερίδια των αγορών που κατακτούμε. Πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό είναι το θέμα του προπολογισμού και επιμένω σε αυτό. Ε, είμαστε φοβερά υποχρηματοδοτούμενοι, ζητήσαμε 35 άτομα προσωπικό και 5 εκατομμύρια ακόμα, μόνο και μόνο για να κάνουμε τα απολύτω απαραίτητα. Ζητώ την ε, υποστήριξή σας. Πώς θα αντιλαμβάνεστε, τα συστήματα τηλεπικοινωνιών βρίσκονται σε οτιδήποτε κάνουμε. Ε, χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μια σταθερή αύξηση στο προσωπικό των προπολογισμό μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προσωπικό, ε, για παράδειγμα, για το ίντερνετ των πραγμάτων, που είναι όλοι νομίζουν ότι είναι μια τεχνολογία του αύριο. Όχι, είναι τεχνολογία του σήμερα. Ήδη εφαρμόζουμε και χρησιμοποιούμε το ίντερνετ των πραγμάτων στα σπίτια μας, σήμερα, εδώ και τώρα. Οπότε χρειαζόμαστε πόρους, χρειαζόμαστε προσωπικό για να εξετάσουμε και αυτό. Δεν λέω ότι μόνο εμείς δουλεύουμε σε αυτό, αλλά έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Κύριε Φρόιντ, Συμφωνώ με τη Χέλη. Το ε, βιβλίο ε, είναι υπερβολικά λεπτομερές και με ένα σενάριο το οποίο δεν είναι πολύ ρεαλιστικό. Ε, μόνο αν γίνει μια φυσική επίθεση, όχι επίθεση στον κυβερνό χώρο, φυσική επίθεση που θα καταστρέψει το υλικό, μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοιου είδου σενάριο. Τις στις περισσότερες φορές, σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων, ε, η επιστροφή στην ομαλότητα θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Αλλά και 24 ώρες να καθυστερήσουμε βέβαια, η ζημιά μπορεί να είναι τεράστια. Ε, όλα αυτά βέβαια διότι είναι, οι επιθέσεις είναι εύκολες και η άμυνα είναι δύσκολη. Και όταν μιλούμε για ασφάλεια, η καλή ασφάλεια συνδυάζει ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία. Αν δεν έχετε και τα τρία συστατικά, να εργάζονται σωστά και με συνεργασία δεν καταλήγεται σε σωστές λύσεις. Οπότε χρειάζεστε τεχνολογία, διαδικασίες και ανθρώπους εκπαιδευμένους. Ο κ. Γιούρι, ε, μίλησε για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Έχουν γίνει τρομοκρατικές επιθέσεις. Ε, για παράδειγμα στο Stuxnet και πάλι οδήγησε σε αλλαγές στην ασφάλεια γιατί μέχρι τότε μιλούσαμε για απώλεια ε, χρημάτων. Όταν συνέβη αυτή η επίθεση μιλούσαμε και, ε, αρχίσαμε να μιλάμε και για απώλεια ζώων. Από τότε αρχίσαμε να εστιάζουμε περισσότερο σε τέτοιου είδους συστήματα ε, και πώς μπορούμε να τα ανακτήσουμε. Οι τεχνικές υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά δυστυχώς είναι δαπανηρές, δαπανηρή εφαρμογή τους. Προσπαθούμε να βρούμε ε, την βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα σε ομαλότητα και οικονομική πραγματικότητα. Και στην Βόρεια Σκανδιναβία είχαμε κάτι παρόμοιο, χωρίς όμως απώλεια ζώων. Ε, Παρ' όλα αυτά τα στήματα θέρμανσης έσβησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα μπορούσαμε να έχουμε απώλεια ζώων εκεί. Κάτι άλλο που συζητάμε είναι μία, ε, μία ενδεχομένως μία ανάλυση, γεωπολιτική ανάλυση κινδύνων. Ε, ορισμένα από αυτά τα οποία είναι απειλές θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τα προβλέψουμε κάνοντας μια γεωπολιτική ανάλυση. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν εντάσεις ή πολύ φτώχεια κλπ. μπορεί να παίρνουν περισσότερες απειλές κλπ. Ενδεχομένως αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε με τους συνεργάτες μας. Μια τέτοιου είδους γεωπολιτική ανάλυση. Αυτά νομίζω. Η πρόεδρος μίλησε, έκανε μια ερώτηση για το διεθνές δίκαιο, αλλά νομίζω το απαντήσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ κύριε Λιφλέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπόθηκαν πολλά, οπότε κάποιες αποχρώσεις θα δώσω εγώ, γιατί σε γενικό βαθμό συμφωνώ με τους προλαλήσαντες, τον Στίβεν και τη Χέλη. Όσον αφορά την έλλειψη πόρων, πρώτα απ' όλα. ασχολούμαστε με πάνω από 61 χώρες ανά τον κόσμο καθημερινά. Και είναι εύκολο να καθορίσουμε από κοινού μια στρατηγική. Το πιο δύσκολο είναι η εφαρμογή της. Και ακριβώ η απειλή στο κυβερνοχώρο είναι κάτι αόριστο, αφηρημένο. Όταν πρόκειται για μια φυσική απειλή, την ξέρετε πότε την έχετε και πότε δεν την έχετε. Ενώ ο ηλεκτρονικός πόλεμος είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει κανείς. Οπότε είναι πιο δύσκολη η απάντηση. Όταν μιλάω με αξιωματούχους υψηλού επίπεδου στις χώρες μέλη, όπως σας είπα, πρόκειται για μια αφηρημένη απειλή, έτσι, και δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι μέρος του προβλήματος του γιατί με τα χρήματα που έχουμε δεν καταφέρνουμε να κάνουμε αυτά που θα θέλαμε. Βέβαια, καταλήγουμε στο να πρέπει να έχουμε ένα συμβάν, να έχουμε μια αποτυχία και τότε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε. Βέβαια, πολλά έχουν να κάνουν αυτό τον εικονικό κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο ο καθένας τον αντιλαμβάνεται. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε τη αυτοκίνητα. Είναι κάτι πολύ πιο αφηρημένο. Όλοι το ξέρουν αυτό, ότι δεν πρόκειται μόνο για την τεχνολογία εδώ, πρόκειται και για την πολιτική που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Τώρα και αυτό που είπατε για τις τρεις εβδομάδες, ε, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά όταν εμείς το κοιτάμε, δεν το βλέπουμε τόσο διαφορετικά από ό,τι ακούσαμε εδώ σήμερα. Δηλαδή, ο κυβερνοχώρος σίγουρα είναι ένα περίεργο μέσο. Πραγματικά χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό, όπως λέμε. Δηλαδή χρειάζεται ένας ε, επιτιθέμενος και ένας στον οποίο επιτίθεται. Δηλαδή εξαρτάται από το πόσο ευάλωτοι είμαστε για να ξέρουμε και τι επίθεση θα δεχτούμε. Άρα εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να δεχτούμε την επίθεση ανάλογα με το πόσο καλά προστατευμένοι είμαστε. Άρα πρέπει να αξιολογήσουμε την ευρύτερη εργαλειοθήκη που μπορεί να διαθέτουμε. Πάντως δεν έχει γραφτεί ακόμα η ιστορία του κυβερνοχώρου. Υπάρχει το IoT, σίγουρα υπάρχουν νέα στοιχεία που καθιστούν ευάλωτο το κυβερνοχώρο, αλλά εγώ τον βλέπω σαν κάτι που περισσότερο μας εξυπηρετεί να κάνουμε πράγματα. Τώρα για τις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Πράγματι, έχουμε διαβάσει πολλά και New York Times λένε ότι θέλανε σε κάποιο ε, το φράχτη να επιτεθούν στη Νέα Υόρκη οι τρομοκράτες. Έχουν δημοσιευτεί πολλά. Όντως υπάρχουν οι ασύμετροι παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτή την τεχνολογία. Φυσικά πρέπει να δούμε πόσο μακριά θέλουν να πάνε. Και πολλές φορές είναι πιο φτηνό και πιο απλό να νοικιάσουν κάποιον ε, βομβιστή παρά να κατασκευάσουν ε, όπλα. Οπότε νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με την οικονομία βάση της οποίας λειτουργούν τέτοια τρομοκρατικά δίκτυα. Και για το κατά πόσο εφαρμόζεται το διεθνές ε, δίκαιο στις ασύμετρες αυτές καταστάσεις, το διεθνές δίκαιο έχει να κάνει με κράτη και όχι με παράγοντες εκτός κρατικής δικαιοδοσίας. Μιλάμε για τις ευθύνες κρατών. Αλλά αυτό ακριβώ είναι που κάνει ο ηλεκτρικός πόλεμος, είναι ότι παρακάμπτει τις δραστηριότητες των χωρών. Υπάρχουν τα άρθρα 5 και 4 όπως γνωρίζετε. Αυτά. Πρόεδρος. Δεν ε, βλέπουμε να ζητάει κάποιος το λόγο. Να κάνω μια παρατήρηση για ένα από τα πράγματα που είπε ε, η κυρία Τίρμα Κλάρα όσον αφορά την οργάνωση της ε, Σανγκάης και την ε, διακήρυξη ε, με τον κώδικα διοντολογίας για τον κυβερνοχώρο. Από τη δική μου εμπειρία είναι λίγο αστείο διότι βασιστών στατιστικών στοιχείων οι περισσότερες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο που προέρχονται από κράτη ε, προέρχονται ε, χονδρικά από αυτή την περιοχή. Ε, ποιες είναι οι εξελίξεις μετά από αυτή την διακήρυξη με τον κώδικα διαντολογίας. Μπορώ να σας εξηγήσω πώς γεννήθηκε αυτή η προσπάθεια. Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο λέγεται διαδικτυακή διακυβέρνηση. Είναι ένα φλέγον ζήτημα αυτή τη στιγμή για ολόκληρη την κοινότητα του κυβερνοχώρου. Πρόκειται για ένα τεχνικό τομέα με πολλά ακρόνημα. Για τον ε, μη εξειδικευμένο είναι δύσκολο να καταλάβει τι συμβαίνει εκεί. Να το εξηγήσω. Κοιτάξτε, το διαδίκτυο δεν ανοίξε κάποια κυβέρνηση, ούτε το διαχειρίζεται κάποια κυβέρνηση, το διαχειρίζονται οι τεχνικέ κοινότητε. Είναι αύλαβη η ε, τεχνική αυτή και αυτοί δημιούργησαν τα δίκτυα αυτή ε, στην Καλιφόρνια για παράδειγμα και αυτοί τα διαχειρίζονται. Είναι ο πρώτος ε, παγκόσμιος τομέας που δεν κυβερνάται από κάποια κυβέρνηση. Ε, μπορεί να εκπροσωπούνται οι κυβερνήσεις σε συμβουλευτικές ομάδες ε, και να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο αλλά η εξουσία τους ε, δεν διαφέρει από αυτή της κοινωνίας των πολιτών ή των τεχνικών. Αυτό είναι, κάτι, είναι μια νέα μορφή διακυβέρνησης. Οι δημοκρατικές χώρες είναι ικανοποιημένε με αυτό, διότι θεωρούμε ότι ο ιδιωτικό κώδικας γράφει καλύτερο κώδικα από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το ίδιο και συμβαίνει και με τα πρωτόκολλα του ίντερνετ. Δεν έχουμε δίποτε πρωτόκολλα ίντερνετ να αξιόπιστα να βγαίνουν από κυβερνήσεις, από κρατικούς μηχανισμούς. Ο ιδιωτικό τομέας ε, είναι αυτός που κυριαρχεί σε αυτόν τον τομέα. Οπότε εγώ θέλω να υπερασπιστώ αυτό το, αυτό το μοντέλο ε, ιδιωτικής ε, διακυβέρνησης του διαδικτύου από τον ιδιωτικό τομέα. Και δεν μπορούν και οι κυβερνήσεις να πούν ε, στον ιδιωτικό τομέα πώς να γράψει κώδικα Ωστόσο, πολλέ κυβερνήσει θεωρούν ότι το διαδίκτυο αποτελεί απειλή για το καθεστώς τους. Και το θέμα με τον κώδικα είναι ότι προσπαθεί να αιτιολογήσει μέσω κάποιες διεθνού συνθήκη συμφωνίας το κυβερνητικό έλεγχο του διαδικτύου. Διότι ο κώδικας ο τελευταίος περιλαμβάνει την παραγραφό 8 που αναφέρεται ότι η κυβέρνηση, το κράτο δεν θυμάμαι ακριβώ διατύπωση, το κράτος θα πρέπει να έχει τον έλεγχο του διαδικτύου. Και αυτό είναι το βασικό κίνητρο για αυτούς τις προτάσεις. Υπάρχουν και άλλα κίνητρα φυσικά, αλλά όπως είδαμε πιο συγκεκριμένα στην Κίνα, έτσι όπως το καθεστώς γίνεται όλο και πιο αυστηρό και περιορίζει την ελευθερία έκφρασης ε, στο διαδίκτυο, διότι ναι, εντάξει, υπάρχει ακόμα κάποια δυνατότητα ελευθερίας έκφρασης, ε, επίκρισης του καθεστώτος και αποφυγής της λογοκρισίας. Ε, ε, είναι κάτι που γίνεται πιο εύκολα στο διαδίκτυο. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μείζον ζήτημα για μας να δούμε κατά πόσο εκεί το διαδίκτυο θα επιβιώσει, διότι η πίεση από πολλές κυβερνήσεις είναι υπαρκτή. Από τότε που το διαδίκτυο μετατράπει σε ένα κρίσιμο πόρο, ζωτική υποδομή για πολλές άλλες ε, επιχειρηματικέ δραστηριότητε, ε, την ηλεκτρονική οικονομία κτλ. Οπότε δεν είναι μόνο για υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου που κάνουμε όλε αυτέ τις προσπάθειε. Υπάρχουν διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος, ε, διάφορα λόμπι, υπάρχουν κίνητρα κατασκοπίας, πολλά διαφορετικά κίνητρα Γι' αυτό οι περισσότερες κυβερνήσεις απαιτούν κάπως περισσότερο κρατικό έλεγχο του διαδικτύου. Και δεν ξέρω τι θα απογίνει με το ελεύθερο διαδικτύο και ποιο θα είναι το μέλλον του. Κατά πόσο θα συνεχίσουμε να έχουμε ένα διελειτουργικό διαδικτύο όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, αν θα έχουμε ένα κατακρεματισμένο διαδικτύο, κατά πόσο θα κατακρεματιστεί σε 4-5 κομμάτια, τα οποία δεν θα συνομιλούν εύκολα, διότι τα πρωτόκολλα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα διαφέρουν. Πιστεύω ότι το μείζον ερώτημα για το τι γίνεται με τη διακυβέρνηση του διαδικτύου ε, παραμένει σε κρεμότητα. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα πρέπει επίση να καταλάβει καλύτερα και αυτά τα ζητήματα τη ε, διαδικτυακή διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ελπίζω να απάντησα. Ναι, βεβαίω. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα την απάντησή σα. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους, ε, τα εξαίρετα μέλη του πάνελ για τη συμβολή τους. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση αυτή. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Δεν είναι απλά ενδιαφέρουσα, αλλά είναι και πολύ σημαντική για ε, τη συμβολή της, τη συμβολή του στη συνολική μας ασφάλεια. Επιπλέον θεωρώ ότι αυτή η διασύνδεση μεταξύ του μη στρατιωτικού και του στρατιωτικού σκέλους είναι ύψης της σημασίας και υψηλής αναγκαιότητας. Οπότε υπολογίζουμε και σε περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στον τομέα αυτών. Ευχαριστούμε πολύ. Να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο που απομένει είναι τα διάφορα, αλλά πρώτα απ' όλα να αποχαιρετήσω τα μέλη του πάνελ και μετά θα συνεχίσουμε.